Dear Καθίστε παρακαλώ. Ξεκινάμε τη συνεδρίασή μας με την έγκριση της ημέρησης διάταξης. Σας ευχαριστώ για την έγκριση. Έχουμε την έγκριση των πρακτικών της 7ης, 9ης, 11ης, 25 και 26 Απριλίου, εάν δεν έχετε αντιρρήσεις έχουν εγκριθεί και αυτά. ανακοινώσει Προέδρου. Υπήρξε συμφωνία στον τριγωνικό διάλογο για την ΜΥΦΙΤ και ΜΥΦΙΡ σε μία μονάχα συνάντηση τριλόγου στις 2 Μαΐου, οπότε η αναδιαβούλευση της Επιτροπής μας με ένα συμπεφωνημένο κείμενο θα λάβει χώρα αύριο. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή και την ομάδα διαπραγμάτευσης για το μεγάλο αυτό επίτευγμα γιατί εξασφαλίσαμε όχι μονάχα την ε, προσαρμογή των ημερομηνιών, αλλά και την ε, προσαρμογή της, της συμφωνία για τη ΜΥΦΙΤ και τη ΜΥΦΙΡ και καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι καθόλου δύσκολο γιατί είναι πολύ δύσκολο να υπάρξουν αλλαγές σε αυτά τα νομοθετήματα, αλλά εμεί το πετύχαμε σε ένα μονάχα τριγωνικό διάλογο με την εξασφάλιση των θέσεων του Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές από το Συμβούλιο. Δεύτερον, να σας πληροφορήσω ότι έχουμε μία νέα επιγραμμική υπηρεσία για όλα τα νομοθετικά, τα νομοθετικά κείμενα που μας δίνει η Διεύθυνση νομοθετικών, Νομοθετικής Παρακολούθησης. Μπορούν να δοθούν λοιπόν προσωπική ηλεκτρονική βοηθή για να μπορούν να παρακολουθούν οι βουλευτές τα στοιχεία αυτά και τις ε, τροπολογίες οι οποίες ε, υποβάλλονται. Η Γραμματεία θα σας στείλει ένα σύνδεσμο για μια σύντομη παρουσίαση αυτού του συστήματος μετά τη συνεδρίασή μας. Συνάντηση συντονιστών. Δύο ορισμοί εισηγητών. Η έκθεση για ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη ειδικών δραστηριοτήτων στον τομέα του, <clears throat> των αναφορών για τα χρηματοπιστωτικά θέματα πηγαίνει στο ΕΛΚ. Η έκθεση για το πρωτόκολλο στη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και του πριγκιπάτου του Μονακό για ισοδύνημα μέσα αυτά της οδηγίας 48 κάθος 2003 έχει συμφωνηθεί επίσης η γνωμοδότηση για την πρόταση για κανονισμό σε σχέση με την δημιουργία ενός προγράμματος διαρθωτικών ε, μεταρρυθμίσεων πηγαίνει στους σοσιαλιστές και επίσης έχουμε αποφασίσει να κάνουμε μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλία για τις ε, εταιρείε FinTech και επίσης μια έκθεση για τα καλυπτόμενα ομόλογα, η οποία θα γίνει αργότερα ο διορισμός. 28 Σεπτεμβρίου θα κάνουμε μια πρόσθετη συνεδρίαση 3 με 5 το απόγευμα με παρουσία εκπροσώπων 28 Μαΐου, συγγνώμη, εκπρόσωπους των Εθνικών Κοινοβουλίων και επίσης μια ανοιχτή συνεδρίαση συντονιστών στις 28 Σεπτεμβρίου με τον κυβερνήτη της, της Τράπεζας της Γαλλίας, τον Φρανσουά Βιλερουά Ντεγκαγιού. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 4 της Ιδέας, κανόνες κατά των πρακτικών φόρο αποφυγής που έχουν άμεσο αποτέλεσμα στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η οδηγία λοιπόν για την αποφυγή της, για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής. Ο κύριος Μπαγί έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Θα συζητήσουμε αγαπητοί συνάδελφοι στοιχείο του φόρου επιχειρήσεων. Αυτό μειώνει σημαντικά τη δυνατότητα των κρατών μελών μας να επενδύσουν, να αντιμετωπίσουν την ένδυα, την, να προωθήσουν την απασχόληση, να βοηθήσουν τα συστήματα υγείας και παιδείας προς όφελος των συμπολιτών μας. Επίσης, είναι φανερό ότι η ενιαία αγορά θα πρέπει να περάσει από μια εναρμόνιση φορολογία των επιχειρήσεων που να είναι ισοδίκαια και αποτελεσματική και θα πρέπει να αποτελέσει ένα από του ακρογωνίου Λίθου τη ενιαία αγορά ο στόχο μα δεν είναι να θίξουμε την οικονομία, αλλά να αντιμετωπίσουμε τα κενά και τι ελλείψει για να υπάρχει ισότητα ανταγωνισμού των επιχειρήσεων και να αποφύγουμε τα σκάνδαλα που έχουμε γνωρίσει πρόσφατα. Η έκθεση αυτή έχει πολλά σημαντικά στοιχεία, τα οποία είναι ακόμα αντικείμενο συζήτηση. Ξέρετε ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε διαφορετικέ πολιτικέ απόψει. Ε, θέλουμε να αποφύγουμε για αύριο το πρωί τι ε, ονομαστικέ κλήσει τη ψηφοφορία, αν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ε, συμφωνίες. Η βασική μας αρχή είναι ότι οι πρέπει να πληρώνουν φόρο εκεί όπου δημιουργούν τα κέρδη τους και γι' αυτό έχουμε μία σειρά από ορισμούς που θα πρέπει να εδραιώσουμε με τα σκάνδαλα αυτά τα, της LuxLeaks και τα λοιπά. Είναι φανερό ότι μεταφέρουν οι πολυεθνικές τα κέρδη τους σε φορολογικούς παραδείσους για να μην πληρώνουν καθόλου φόρους. Σε ό,τι αφορά τώρα την ε, εξαίρεση από τη φορολογία των τοκοχρεολησίων η Κομισιόν έχει ε, μια θέση που το Κοινοβούλιο θέλει να την τροποποιήσει με ένα μέγιστο ποσοστό 10% για την, αφαίρεση αυτή. Και επίσης ε, θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο θα επιτρέψει στις πολυεθνικές οι οποίες δεν προβαίνουν σε πόρο αποφυγή να χρησιμοποιήσουν αυτή τη δικλίδα της μη φορολόγησης των τοκοχρεωλησίων. Επίσης είναι σημαντικό για τις ε, επιχειρήσεις οι οποίες ε, δεν χρησιμοποιούν τα συστήματα φοροαποφυγής να έχουν ε, μια ορθή μεταχείριση και επίσης θα πρέπει να υπάρξει ένας κατάλογος των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν φορολογικούς παραδείσους. Επίσης, οι επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας με τεχνητό τρόπο για να μειώσουμε <clears throat> τα κέρδη τα οποία δηλώνονται. Αυτό είναι σε βάρος των χωρών οι οποίες δημιουργούν καινοτομία και θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει μια ελάχιστη ε, φορολόγηση ώστε να ευνοηθεί η τεχνολογική πρόοδος. Ένα άλλο σημείο. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει μια ε, εισοδή και φορολογία των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν οι, τα κράτη-μέλη να επιβάλλουν εθνικού φόρου στα κέρδη πολυεθνικών συναδελφών του που φορολογούνται με λιγότερο από 15% σε άλλε χώρε. Αυτό θα είναι ένα στοιχείο αντιμετώπιση τη φοροαποφυγή. Γιατί αν δεχτούμε την πρόταση τη Κομισιόν να υπάρχει ένα ποσοστό διακειμενόμενο 40% του ε, της ελληνικής φορολογίας. Αυτό θα οδηγήσει σε μεγάλες ε, διαφορές μεταξύ των χωρών, γιατί στη Βουλγαρία είναι 4% η φορολογία των επιχειρήσεων, 12% στη Γερμανία. Τέλος, ε, έχουμε μία πρόταση για την εναρμονισμένη κοινή βάση για την φορολογία των επιχειρήσεων και μια κοινή θηρίδα για την υποβολή των ε, δηλώσεων αυτών για τη φορολογία ώστε να εξασφαλίσουμε την ε, διαφάνεια. Ξέρω ότι είναι μια πολύπλοκη έκθεση με πολλές ε, διαφωνίες σε πολιτικό επίπεδο. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε αύριο μια, μια ε, ισχυρή πλειοψηφία για να καταδείξουμε ότι εμείς θέλουμε να υποστηρίξουμε τον αγώνα κατά της φοροφυγής. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές οι οποίοι έχουν λάβει μέρος στην διαβούλευση για τα θέματα αυτά. Σέβομαι πάρα πολύ το έργο του και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε αύριο να καταλήξουμε σε μια θετική ψηφοφορία. Thank you to the Ευχαριστούμε πολύ τον εισηγητή και τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Νίτερ Μάγερ για το ΕΛΚ. Thank you very much, Mr. Chair. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Έχω ορισμένε παρατηρήσει. Δεν μπορώ όμω να σα πω την τελική τοποθέτησή μα πρώτα-πρώτα, γιατί έχουμε μια συνάντηση το απόγευμα και μόλις πριν από λίγα λεπτά πήρα την ε, νεότερη ε, εκδοχή των ε, συμβασικών τροπολογιών. Κάπως εξεπλάγει από το πώς έχουμε χειριστεί το θέμα, διότι από ό,τι φαίνεται με αυτή την έκθεση θέλουμε να υπάρξει η με και με πράσινους μια συνένεση ε, όμως δεν υπάρχει για τόσο σημαντική έκθεση ε, τελικά με αυτούς τόσο μεγάλη σύνεση. Νομίζω ότι θα πρέπει να αποδείξουμε ότι είναι ενωμένο εν προκειμένου το Κοινοβούλιο. Τέλος πάντων από τότε που άρχισε η διαδρομή αυτής της έκθεσης. Εγώ έχω βοηθήσει τον εισηγητή, του έχω παράσχει κάθε φορά το πληροφορίε τις πληροφορίες του ποιες είναι οι μας. Δεν ε, είναι και μεγάλη συζήτηση, ε, γιατί έχουμε κάποια σημαντικά σημεία που θέλαμε να προβάλλουμε και δεν ελήφθησαν υπόψη για την ε, φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή, για κάποιες αθέμητες πρακτικές. Όλα αυτά είναι πολλές προτεραιότητες για μας. Θα πρέπει επίσης να μην κατέβουμε σε μια οδηγία που να σκοτώνει τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την ε, φορολογία κάποιων επιχειρήσεων, τα οι οποίες δεν ε, κάνουν ζαβολιές, αυτό κατά κάποιο τρόπο να μην τις τιμωρήσουμε και έχουμε προτείνει σχετικά. Αυτός είναι και ο σκοπός μου εδώ ε, να υπάρχει επίσης κάποιο είδους τεχνική τεκμηρίωση για κάποια σημεία της ε, οδηγίας. Ε, ζητήσαμε τη γνώμη των άλλων, δεν μας είπαν τίποτα. Τώρα έχουμε, έχουμε ε, στο A, B μέχρι το H κάποια προβλήματα και κάποιες συνεργασίες προβλίες. Για το FG επίσης θα πρέπει να δούμε τι οριακές τιμές θα καθοριστούν και θα πρέπει να δούμε τι κανόνες, τι κριτήρια θα θεσπιστούν, θα υπάρχουν ε, εθνικές ρυθμίσεις ε, ή υπερεθνικές. Εγώ θα έλεγα για το ποσοστό να έχουμε σαν κατόφλι 25%. Το ποσοστό πάνω από το οποίο δηλαδή θα αυξάνεται η φορολόγηση. Πάντως, το κλειδί είναι η συμβαστική B το θέμα του περιορισμού των επιτοκίων. Interest limitation. Αυτό να προσέξουμε επίσης, να δούμε τι θα γίνει με την Επιτροπή αλλά και με το Συμβούλιο γιατί ε, δεν ισχύει το ότι του 30% κάτι θα αλλάξει. Έχουμε και την έκθεση του ΣΑΠ που λέει ότι έχουμε μέχρι 38%. ότι δεν θα είναι δυνατόν να εκπέσει κάποιες δαπάνες από τη φορολογική αίλια. Και βέβαια κάποιοι θα πληρώσουν παραπάνω και κάποιοι πρόκειται να αποφύγουν τη φορολογία. Αλλά σύμφωνα με τον ΑΣΑ, το ποσοστό που ισχύει είναι το 13% και αυτό μου φαίνεται αρκετό, αλλά τουλάχιστον είναι λογικότερο. Κάτι άλλο πρέπει να λάβουμε υπόψη στην Ευρώπη. Έχουμε μεγαλύτερη αναλογία δανείων για εξυπηρέτηση και χρηματοδότηση των εταιριών για τις επενδύσεις τους. Οι δύο σημείμοι ε αυτό κάνουν. Επεκτείνουν τις εργασίες τους με χρηματοδότηση, με πίστοση. Άρα θα πρέπει κάτι να γίνει με αυτό το επιτόκιο που λέει το κείμενο. Θα έχουμε με αυτά τα οποία προτείνονται μεγάλη περιστολή του περιθωρίου κέρδους και αυτό το κατόφλι του 10% σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουν να επικαλεστούν το επιτόκιο οι εταιρείε για φορολογικού σκόπους. Επίσης, άλλο πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε και τις χώρες της Ευρωζώνης που τουλάχιστον προς το παρόν έχουν αρκετά χαμηλά επιτόκια και επιβάρυνση όσον αφορά το επιτόκιο για τις ε, εταιρείε με καλή επίδοση. Όμως, εκτός Ευρωζώνης, ας πούμε στην Ρουμανία, τελευταία δεκαετία, κάθε χρόνο έχουμε αύξηση κατά 20% της χρηματοδότησης. Το 2010 είχαμε 40%. Το 2013 είχαμε το επιτόκιο πάνω από 10%. Όμως, πώς θα καλυφθούν αυτές οι χώρες ε, αν έχουμε κατόφυλλο τόσο χαμηλό. Και έχουμε επίσης το διατραπεζικό επιτόκιο στην Πολωνία που είναι πάνω από 6% τη σημερινή μέρα. Γι' αυτό και σας λέω. Θα πρέπει να λεφθεί υπόψη το τι ισχύει για τις επιχειρήσεις. Πώς θα ωφελήσουμε την οικονομία. Γι' αυτό λέω και εγώ ότι αυτά τα οποία ο εισηγητής προτείνει δεν με βρίσκω σύμφωνο και θα εισηγηθώ να καταψηφίσει την πολιτική μου. Point of order. Yes. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να μιλήσω γερμανικά. Κύριε Πρόεδρε, άκουσα τον συγητή ότι δεν υπάρχει ακόμα συνεννόηση μεταξύ των μεγάλων ομάδων και θα υπάρξει διαπραγμάτευση απόψε για το αν ε, μπορούμε να έχουμε ευρύτερη πλειοψηφία στην Επιτροπή και άρα από ό,τι φαίνεται οι συμβαστικές προτάσεις ε, που υπάρχουν τώρα επιτάπιος θα, έχουν, θα αποκτήσουν νέα μορφή. Ε, δεν μπορούμε έτσι να ψηφίσουμε όμως αν αλλάξουν απόψε οι συμβαστικές προτάσεις. Είναι δύσκολη, περίπλοκη έκθεση και πρέπει οι βουλευτές να προλάβουν να τις διαβάσουν τουλάχιστον. Άμα τις λάβουμε απόψε, με στη νύχτα ή αύριο το πρωί και όλας, ε, πώς θα δουλέψουμε. Γι' αυτό ζητάω να αναβληθεί η ψηφοφορία για να έχουν την ευκαιρία τουλάχιστον να το διαβάσουν οι βουλευτές. Να διαβάσουν τι θα ψηφίσουν. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, έχει εγκριθεί η ημερήσια διάταξη, τώρα δεν αλλάζει. Και είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό το κοινοβούλιο να τοποθετηθεί πριν από το ΕΚΟΦΗΝ. Πρέπει να λάβουμε και αυτόν υπόψη. Αυτό. Α, βεβαίως, εντάξει, αντιλαμβανόμαστε την συζήτηση εντό των ομάδων και από όσο καταλαβαίνω υπάρχουν μία-δύο ακόμα συμβιβαστικές που είναι αντικείμενο διαπραγματεύσεων. Οι περισσότερες ε, ισχύουν. Και λογικό είναι κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης να αλλάξουν κάποιες λεπτομέρειες εάν αυτό χρειάζεται. Προσωπικά λοιπόν δεν θα ακολουθήσω την συμβουλή σας γιατί νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό το Κοινοβούλιο να τοποθετηθεί. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση. Εγκρίναμε λοιπόν την ημερήσια διάταξη. Τώρα θα γίνει μια συζήτηση. Δεν ξέρω ποια θα είναι η άποψη ε, και του εισηγητή. Οπότε ήταν και πολύ αργά και πολύ νωρίς αυτό το οποίο είπατε γιατί ήταν ε, αφού ορίστηκε η ημερήσια διάταξη και πλέον ολοκληρωθεί η συζήτηση. Θα παραμείνει λοιπόν η ημερήσια διάταξη. Κύριε Λάγγεν. Ναι, εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με τον κύριο Λούκε. Δεν είναι δυνατόν εμείς να στυλώνουμε τα πόδια και να λέμε θα ψηφίσουμε χωρίς να ξέρουμε μετά την πράσινη εβδομάδα κιόλα τι μορφή θα έχουν ε, οι συμβαστικές προτάσεις. Είναι μονομερής και λανθασμένη η πρότασή σας. Πρέπει να ψηφίσει ολόκληρη η Επιτροπή νομίζω. Thank you, Mr. Lange, um, σας ευχαριστώ κύριε Λάγκεν. Και ε, παράξενο θα ήταν να γίνει συζήτηση τη μέρα πριν από την ψηφοφορία. Ποιο το νόημα της συζήτησης σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή έπρεπε να τα έχουμε αποφασίσει όλα εκ των προτέρων. Θα μπορούσαμε να καταργήσουμε και τη συζήτηση πριν από την ψηφοφορία, άμα είναι έτσι. Η συζήτηση επίσης έχει το νόημα του να πείσει ο ένας τον άλλον, αλλιώς θα είναι άχρηστη. Οπότε προτείνω να κλείσει αυτή η συζήτηση και μετά θα δούμε αν προτείνει κάτι ο εισηγητής και θα γίνουν οι σχετικές ε, διαβουλεύσεις. Ε, αυτή τη στιγμή ισχύει η μερίσια διάταξη. Και εγώ επιμένω να είμαστε έτοιμοι για να προλάβουμε τουλάχιστον το Συμβούλιο. Κύριε Μπάλτς. Κοιτάξτε, εγώ έχω καλή διάθεση και στο είμαι χαλαρός ε, μετά από την πράσινη εβδομάδα. Δεν ήθελα να πάρω τον λόγο, αλλά αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Λούικ και ο κύριος Λάγκεν. Αλλά τώρα, αν θέτε να είμαστε τυπικοί, και εσείς ως πρόεδρος δηλαδή, θα ήθελα να υπενθυμίσω πως αποφάσισαν οι συντονιστές ότι μέχρι Δευτέρα 3 η ώρα και τώρα είναι 16 και 18. Εάν μέχρι Δευτέρα 3 η ώρα δεν υπάρχουν ε, συμβαστικές προτάσεις, δεν είναι δυνατή η ψηφοφορία την επομένη. Άμα είναι να είμαστε τυπικοί. Θα ήθελα λοιπόν ως ΕΛΚ να παρακαλέσω να τηρήσουμε τα συμφωνηθέντα. Σας ευχαριστώ. Μπουρκάρτ Από όσο καταλαβαίνω, Έχουμε λάβει το κείμενο πριν τις 3 η ώρα. Βεβαίως. Άρα είμαστε μέσω στους κανόνες. Αν μια πολιτική ομάδα, η δική σας προκειμένου, ζητήσει από τον εισηγητή να τροποποιηθεί η συμβαστική πρόταση και άρα το δεχτεί μετά ο εισηγητή, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί η ομάδα η οποία ζητάει αλλαγή του συμβιβασμού μετά να έρθει να μας πει «Α, όχι, τώρα δεν μπορούμε να ψηφίσουμε». Τα ξαναλέω. Λοιπόν, έχουμε ένα κείμενο συμβαστική πρόταση, το οποίο έχει κατατεθεί εγκαίρω σύμφωνα με τον κανονισμό. Τώρα υπάρχει μια συζήτηση, η οποία δεν έχει λήξει. Οπότε για μένα είναι ε, δύσκολο να λάβω απόφαση στη μέση της συζήτησης. Δεν είναι τέτοιο ζήτημα στην ημερήσια διάταξη πριν από λίγα λεπτά. Ρώτησα, εγκρίναμε ομοφόνο στην ημερήσια διάταξη. Τώρα αλλάξατε άποψη, αλλά Υπάρχει ένα κείμενο που κατετέθη εγκαίρως και εάν έχω καταλάβει σωστά τον κύριο Μάιρ, ένα αίτημα αλλαγής κάποιο πράγματος. Και μετά δεν ξέρω ποια θα είναι η απάντηση του εισηγητή. Ας ολοκληρωθεί η συζήτηση και να λάβουμε την απόφασή μας στο τέλος της συζήτησης. Μέχρι στιγμής έχουμε εγκρίνει μια ημερήσια διάταξη. Πριν από λίγα λεπτά μόλις. Λοιπόν, κύριε Λούνες για το σημείο αυτό και μετά θέλω να αναφερθώ ως χειώδης συζήτης. Θέλω να επιμείνω σε αυτό που είπε ο κύριος Λούκε και ο κύριος Μπάλτς ως Εμείς θεωρούμε ότι όλα αυτά τα οποία έχουμε συμβαστικές ε, λύσεις είναι, προβληματικές. Δεν έχουμε μοναχα μία ή δύο Συμβαστικέ να τροποποιήσουμε και τα άλλα θα είναι εύκολα. Όχι, είναι πάρα πολλά τα οποία πρέπει να τροποποιηθούν. Αν αυτό το οποίο θέλει ο εισηγητή να έχουμε μια ευρεία πλειοψηφία μπορεί να επιτευχθεί. Γι' αυτό θέλω να υπογραμμίσω και να υποστηρίξω αυτά που είπε ο κ. Λούκε και ο κ. Μπάλτ. <coughs> Ευχαριστώ. <coughs> Ο κ. Καλβέζο Ζαμπόν έχει το λόγο. Όχι, όχι, αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι της παρέμβασής μου επί της ημερήσιας διάταξης. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα νομίζω πως ε, και η αίσθηση στην αίθουσα είναι πως η αρχική πρόταση της ε, Κομισιόν ήταν ε, ήδη αμφίβολη και πλέον έχει αμφισβητηθεί ε, και από τα αριστερά κόμματα και δεν είναι πλέον κατά του ΜΠΕΦΣ αλλά είναι κατά των επιχειρήσεων και τα αριστερά κόμματα θα έπρεπε νομίζω να έχουν την ειλικρίνεια να μας πούν ποια είναι τα κίνητρά τους. Το θέμα δεν είναι να καταπολεμήσουμε τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές αλλά να τιμωρήσουμε όλες τις επιχειρήσεις τελεία. Αν θεωρείτε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι νησί και δεν επηρεάζεται από τον υπόλοιπο κόσμο και δεν πρέπει να ενισχύσουμε την ε, ελκυστικότητά μας, απλά πείτε το. Αν ε, θέλετε να τρέχουμε πίσω από τα μεγάλα κράτη-μέλη, πείτε το. Γιατί όπως και ο κύριος Νίτερμαϊερ έτσι και εγώ ανησυχώ για την κατεύθυνση την οποία παίρνουμε. Οπότε σας παρακαλώ ας επιστρέψουμε στην ουσία της ε, συζήτησης και ποια είναι η ουσία της ε, συζήτησης και θα το τονίσω η καταπολέμηση της φοροαποφυγής, το επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού είναι πρώτη προτεραιότητα. Αυτή είναι η άποψη του ECR και χαίρομαι που τα κράτη-μέλη υποσχέθηκαν ότι θα επιβάλλουν τα μέτρα της τελικής έκθεσης του BEPS. Το μάθαμε αυτό και από την συζήτηση περί Πάναμα ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε τη φοροαποφυγή και αν ήταν όλοι οι ειλικρινείς ε, θα μπορούσαν να κατέβουν οι φόροι. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι νησί, δεν είναι απομονωμένη. Είμαστε σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Διεθνώς ε, γίνονται πάρα πολλές ε, συμφωνίες, σύμφωνα με την πρόταση του USO, και θα πρέπει άρα να πάμε λίγο παραπέρα. Από ό,τι φαίνεται τα μισά από αυτά τα οποία προτείνει η Κομισιόν δεν προέρχονται από το σχέδιο δράσης αυτό και ειλικρινά απογοητεύτηκα λίγο από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί ακριβώς ε, πηγαίνει πολύ περισσότερο από αυτά τα οποία θέλει το USO και ακριβώς αυτό θα βλάψει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών κρατών μελών. Γιατί βλέπουμε πως ο θέλει να πάει ακόμη παραπέρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι ιδέες συμβαστικής σας ε, προτάσεις δεν μου φαίνονται και τόσο συμβαστικές. Μου φαίνεται πως είναι μια σειρά απαιτήσεων από τις ε, πιο αριστερές ομάδες ε, του Κοινοβουλίου αυτού. Παραδείγματο χάρη λέτε πως θα πρέπει να περιοριστεί η έκδοση του φόρου μέχρι το 10%. Αυτό σημαίνει πως 38% των επιχειρήσεων θα πληρώνει περισσότερους φόρους. Αυτό σημαίνει ότι θεωρούμε τι δηλαδή, ότι είναι απαταιώνε σήμερα το 38% των επιχειρήσεων. Α είμαστε λίγο σοβαροί. Θα τιμωρήσουμε τους συνεπεί επιχειρηματίε που πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και ειδικά τους μικρομεσαίους. Τέταρτον. Έχετε εδώ πέρα κάνει μια επιλογή υπέρ των ε, κρατών μελών, των μεγαλύτερων και κατά των μικρότερων όπως το Βέλγιο. Θα βλάψει το Βέλγιο η πρότασή σας. Γιατί βεβαίως ακολουθείτε μία πρόταση ε, για το 30% των ε, καθάριστων κερδών που θα πρέπει να εξαιρείτε και όλο τυχαίως είναι μία πρόταση που έχει κάνει ένα από τα μεγαλύτερα κράτη. και πάλι εδώ πέρα μας λέτε πως θα πρέπει φορολογία να λαμβάνει χώρα εκεί όπου ασχείται η οικονομική δραστηριότητα. Άλλη μία επίδειξη πολιτικής ε, ισχύω. Και τέλος κύριε Πρόεδρε. Έχω την εντύπωση πως ε, με την πρόταση αυτή ε, θα καταλήξουμε σε όλο και υψηλότερους ε, φόρους. Η Κομισιόν λοιπόν έχει ακολουθήσει μια λάθος ε, κατεύθυνση και λάθος για τα μικρότερα κράτη-μέλη. Εκμεταλλεύτηκε το κλίμα αυτό, Σουίς, Λίξ και Παναμά για να αυξήσει τους φόρους, αλλά έτσι θα τιμωρήσει τις ε, επιχειρήσεις που κινούνται καλή τυπιστή. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Και αυτό θα καταλήξει σε λιγότερες επιχειρήσεις και λιγότερες επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα πρέπει τέλος να συζητήσουμε, όταν συζητούσαμε μάλλον το σχέδιο του Γιούνκερ, όλοι λέγαμε το πώς θα γίνει η Ευρώπη πιο φιλική για τις επενδύσεις. Εδώ πέρα κάνουμε ακριβώς το αντίθετο και θα έχουμε λιγότερες θέσεις εργασίας. Πρέπει να αντιληφθούμε το τι ψηφίζουμε. Τα όσα ψηφίζουμε εδώ μέσα τα διαβάζουν και εκτός. Και σβήνει το μικρόφωνο του ομιλητή. Εντάξει, λέει ο πρόεδρος. Καλβέ Σαμπόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από την ομάδα των φιλελευθέρων θα ήθελα να πω, προσπαθώ να είμαι σύντομο. Εμεί προφανώ θέλουμε να δώσουμε ένα στεναρό μήνυμα. Νομίζω ότι το περιμένει όλη η κοινωνία από εμά μετά από τα πρόσφατα γεγονότα και ακόμα και από αυτά τα γεγονότα που ακολούθησαν την πρόταση τη Κομισιόν. Θέλουμε να δώσουμε ένα στεναρό μήνυμα σε ό,τι αφορά το να κλείσουμε τα παραθυράκια τα οποία επιτρέπουν αυτήν την αποφυγή. που δεν είναι ενέργειες οι οποίες είναι παράνομες απλώς είναι η χρησιμοποίηση και η εκμετάλλευση κανόνων που είναι κακώς διατυπωμένοι και πρέπει να το εξασφαλίσουμε ότι θα βελτιωθούν αυτοί οι κανόνες πρέπει να βρούμε τρόπους να έχουμε νέους κανόνες οι οποίοι θα τονίσουν ότι κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός. Επίσης, πρέπει να καταλάβουμε ότι μια ευρεία πλειοψηφία στο κοινοβούλιο μας έχει πρέπει να υποστηρίξει ένα κείμενο αυτού του είδους. Αυτά θέλουμε να υπογραμμίσουμε ως ομάδα της ΑΝΤΕ και αυτός είναι ο στόχος μας. Όπως ξέρουν όλοι, μπορούν να υπάρξουν διαφορετικές ε, ερμηνείες των αριθμητικών στοιχείων, αλλά τελικά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε κάποιες πολιτικές αποφάσεις μέσα στα όρια του ε, λογικού, μέσα στα όρια αυτού που έκανε ο ΩΣΑ. Και η ομάδα μας πάντα θέλει να έχει μεγαλύτερη αυστηρότητα στις ενέργειες του Κοινοβουλίου και θέλει να υποστηρίξει μια συμφωνία μεταξύ των πιο μεγάλων πολιτικών κομμάτων. Υπάρχουν κάποια σημεία που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν και να βρεθούμε μια λύση. Η... Το... Τα ποσά που εκπέ... εκπίπτουν από την εξυπηρέτηση των ε, δανείων. Εμείς είχαμε υποστηρίξει ένα 10% και είπαμε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια ε, παράταση αυτού του καθεστώτος ε, μείωση κατά 10% για πέντε χρόνια, ώστε ορισμένες δράσει επενδυτικέ που έχουν να κάνουν με υποδομές να μπορέσουν να μην θυγούν. Η ομάδα μας θεωρεί ότι το 20% δεν θα δώσει ένα αρκετά ισχυρό μήνυμα. Αλλά με το 20% μπορούμε να φτάσουμε εάν κάποιες μεγάλες πολιτικές ομάδες ενδεχομένως να μπορέσουν να το δεχτούν. Γι' αυτό δεν πρέπει να παραμείνει άκαμπτος ο εισηγητή στο 10% εάν είναι δυνατόν να ευρεθεί με άλλο ποσοστό κάποια συμφωνία. Τώρα, ένα άλλο θέμα, το θέμα των ευρεσιτεχνιών. Ο τρόπος αυτός ο στρεβλός να παρουσιάζονται έτσι οι επενδύσεις. Σίγουρα θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την παραπλανητική λειτουργία του συστήματος, αλλά θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συνδέουμε αυτές τις ε, επενδύσεις στις πραγματικές παραγωγικές ε, ενέργειες των επιχειρήσεων και όχι να γίνεται με ένα παραπληκτικό τρόπο. Αυτό το οποίο δεν θέλουμε να γίνει και δεν είναι χρήσιμο είναι να χρησιμοποιήσουμε όλο αυτό το σύστημα για να καταφερθούμε και πάλι κατά των επιχειρήσεων και να τις επικρίνουμε. Γιατί δεν είναι αυτό το θέμα. Ούτε μπορούμε σε κάποιες ε, αιτιολογικές σκέψεις έστω να πούμε ότι η πρακτική αυτή πρέπει να σταματήσει τώρα μέχρι την τάδε ημερομηνία. Δεν θα πρέπει να είμαστε λοιπόν μεροληπτικοί για τα θέματα αυτά. Γιατί τη ρήτρα switch over επίσης. Μπορούμε να υποστηρίξουμε το 25% εμείς ε, θεωρούμε ότι είναι πιο λογικό να έχουμε μία φορολογία κατά αποκοπή. Αλλά δεν πιστεύω ότι πρέπει να σταματήσουμε την δυνατότητα επίτευξη συμφωνίας γιατί διαφωνούμε μεταξύ του 10% και του 15%. Η Άλτε λοιπόν θέλει την πιο απαιτητική λύση, τουλάχιστον τα περισσότερα μέλη μας αυτό θέλουμε. Εμείς θα θέλουμε όμως πάντα να υπάρξει ένα, μια συμφωνία. Γιατί δεν υπάρχει μαγικό αριθμό. ούτε το 10, ούτε το 15, ούτε το 13, ούτε το 25. Όλα αυτά αλλάζουν από, το χρόνο στο, από χρόνο σε χρόνο. Είναι πολύπλοκη η οικονομία. Δεν θέλω λοιπόν να ε, μακρηγορήσω, φτάνω πια τα 5 λεπτά. Νομίζω όμω ότι υπάρχει δυνατότητα να βρούμε μια συμφωνία, να έχουμε ένα καλό πολιτικό κείμενο το οποίο να συλλέξει την πλειοψηφία των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και σα λέω και πάλι, δεν υπάρχει λόγο να κάνουμε όλα αυτά ένα φιλιππικό κατά των επιχειρήσεων <clears throat> και ούτε θα πρέπει να δώσουμε την ε, εντύπωση ότι αυτό που θέλουμε είναι να πληρώνουν περισσότερο φόρο οι επιχειρήσει. Απλώ θέλουμε να σταματήσει η φοροαποφυγή και αυτοί που φοροαποφεύγουν να πληρώνουν του φόρου που του αναλογούν. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρο, ο Φάμπιο Ντεμάζη, έχει το Ναι, χαιρετίζω το γεγονό ότι έχει συζήτηση τώρα που γίνεται η συζήτηση. Τώρα να σας, πω τη φωνή της λογική σου, τη Γκουε. Να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή, εργάστηκε με άριστο τρόπο και έχουμε πολλούς λόγους και από το Panama και από το LuxLeaks ε, να κάνουμε κάτι για το ξέλιμα χρημάτων γιατί αυτό περιμένει ο κόσμος. Άρα θα πρέπει να ενώσουμε όλες τις προσπαθίες μας και πρόεδρε παρακαλώ να επιβάλλετε λίγη ησυχία στην αίθουσα ή δυνατόν λέει ο κύριος Ντεμάζη Thanks. So, first of all, with all due respect to my colleagues... Με όλο το σεβασμό στους συνέλφους από ECR και EPP θέλω να σας πω το ότι η καταπολέμηση της ε, φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής και ότι αυτό θα σκότωνε τις επιχειρήσεις. Μα δεν καταλαβαίνω. Εσείς τι επιχείρηση έχετε κατά νου όσον αφορά του ομιλου εταιρεών στην Ευρώπη, τα νομικά πρόσωπα στην Ευρώπη, γιατί ε, εδώ πέρα κινήθηκε ο εισηγητή στα όρια του ΟΣΑ. Τα είπαμε και την περασμένη εβδομάδα με του αδέλφους και πολλά από τα σημαντικά σημεία που καλύπτει ο εισηγητής ευθυγραμμίζονται 100% με αυτά τα οποία τώρα κουβεντιάζει η Αμερική. Μα τι, η Αμερική είναι κατά των επιχειρήσεων Ποιος, ποιος είναι το 100 τελικά ή στην Αμερική, είτε και εδώ στην αίθουσα στη δική μας. Οπότε είπαμε ότι θα συμφωνούμε με τον εισηγητή να περιοριστεί στο 10% των κερδών προφόρου το ποσό που εκπίπτει από τα πτώκια. Όμως ακόμα και αν δεν ευθυγραμμιζόμαστε με την Αμερικανική ρύθμιση, ευθυγραμμιζόμαστε με τον ΩΣΑ. Τώρα, για το κατόφλι, 15% συμφωνούμε. Συντελεστής 15% επομένως αυτό να επιβληθεί. Αυτό θα πρέπει να επιβάλλουν και τα κρατημετρό όσον αφορά ε, τις ασυμβατότητες του υβριδικού τύπου θα πρέπει να μην είναι υποχρεωτική για τρίτες χώρες και εμείς είμαστε υπέρ του εξή. να γίνει φορολόγηση στην πηγή. Και αυτό το έχει επισημάνει η Επιτροπή επανειλημμένα. Γιατί σε πολλές χώρες, όπως τις κάτω χώρες, θα πρέπει να σταματήσει η απόκρυψη φορολογητές ύλης σε φορολογικούς παραδείσους. Έχουμε αυτά τα boxes της καινοτομίας. Τα έχουμε πει πανελειμμένα, λαμβάνοντας υπόψη ε, τον Σάκη και στο Παρίσι και συγκλίνουμε τα υπόψη μας με το Υπουργείο των ε, Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν υπάρχουν στοιχεία, ακόμα και η Γερμανία συμφώνησε, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι αυτές οι καινοτομίες πρόκειται να βοηθήσουν ε, την ε, έρευνα. Υπάρχουν καλύτερα εργαλεία. Επίσης, πρέπει να δούμε τι γίνεται με αυτά τα έξοδα για την αδειοδότηση, γιατί τώρα υπάρχουν πολλά περιθώρια για παρατυπίες ακόμα και αν η χώρα του προορισμού δεν φορολογεί θα πρέπει να επιβληθεί ένα όριο όσον αφορά το κατά πόσον εκπίπτονται αυτά τα τέλη ή έξοδα για την έγκριση αδειοδότηση. Είμαστε αποφασισμένοι και αυτό θα πρέπει να δείξουμε ότι θέλουμε να ωφελήσουμε την πλειοψηφία των πολιτών. Να συμπήξουμε κάποιους ε, συμβιβασμούς προς αυτή την κατεύθυνση και για αυτό το λόγο. Άρα θα πρέπει όλες οι πολιτικές ομάδες να αναθεωρήσουν την τοποθέτησή τους ε, κοιτώντας τα μάτια των πολίτη όσον αφορά τα φορολογικά τους συμφέροντα των πολιτών. Ε, η Εύα δεν μπόρεσε να έρθει πρόεδρε και στη θέση θα πω τα εξή. Πρώτα πρώτα σύντομα να σας πω ότι ο σκοπός δεν είναι να αυξηθεί ο εταιρικός ε, φόρος. Ούτε θέλουμε να εμποδίσουμε την οικονομία. Θέλουμε να κλείσουμε κάποια παραθυράκια που τώρα τα εκμεταλλεύονται κάποιες πονηρές εταιρείε. Πραγματικά θεωρώ ότι οι προσπάθειε του Κοινοβουλίου για να υπάρξει συνένεση είναι κάτι ε, πάρα πολύ αξιόλογο. Ε, προσπαθούμε όλοι να συγκλίνουμε και να κάνουμε τη δουλειά μας ως πολιτικοί. Επί της ουσίας τώρα ευχαριστώ τον εισηγητή, όπως παραδοσιακά γίνεται, αλλά ευχαριστώ και τους άλλους ε, σκιώδες το θέμα. Είναι πολύ σημαντικό. Και βασικό στόχο του Κοινοβουλίου είναι να στείλει μήνυμα ξεκάθαρο στο Συμβούλιο γιατί θα πρέπει να είναι η πρόταση φιλόδοξη. Και έτσι να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Να μην αφήσουμε παραθυράκια τα οποία να γίνουν αντικείμενα εκμετάλλευση για τέτοιε κακέ πρακτικέ. Όμω βλέπουμε ότι έχει απονευρωθεί η στάση του Συμβουλίου δυστυχώ. Οπότε και εμεί υπονομευόμαστε. Αλλά σε πολλέ περιπτώσει θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι. Άλλε ε, περιπτώσει θέλουμε να προχωρήσουμε περισσότερο, άρα θα πρέπει να εμείνουμε όσον αφορά τις, ε, τους κανόνες που δίνουν τις ξένες εταιρείες και τελικά να γίνει τη φορολόγηση στη χώρα υποδοχής τη εταιρεία, εκεί που είναι δηλαδή η δραστηριότητα. αυτό το 15% θα πρέπει να ισχύσει και επίσης νομίζω το Κοινοβούλιο θα πρέπει να μείνει σε αυτές τις ασυμβατότητες και να μην έχουμε τι εταιρείε ούτως ώστε να με δημιουργικό τρόπο να κινούνται έτσι ούτως ώστε να μεταβούνται κάποια παράθυρα επίσης το Κοινοβούλιο να είναι αποφασιστικό όσον αφορά την καταπολέμηση αυτών των ε, πρακτικών που θα πρέπει οι δραστηριότητε οι ερευνητικέ να υποστηριχτούν να μην έχουμε και προς αυτή την κατεύθυνση φόρα αποφυγή και να ρυθμίσουμε επίσης ε, τα κατόφλια που προτείνω αυτό που λέει ο ΣΑΟΣ όσον αφορά τα ποσά και τα μεγέθη που εκτύπτουν. Άρα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τη μόνιμη εγκατάσταση. Εμείς επιμένουμε ε, ότι θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει στις φορολογικές ρυθμίσεις, θα πρέπει όλα αυτά να είναι γνωστά, δημοσιευμένα, να δούμε πώς δεν θα υπάρχει κάποιο συμπεγνία με κάποια κρατημέλη ε, και να δούμε τι, τι θα γίνει με τον ορισμό του TST φορολογικός παράδεισος να μην καταλήξουμε σε κάποιες ε, παρεκκλήσεις που θα καλύψουν κάποιες ε, χρηματοοικονομικές συναλλαγές θα πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το καθεστώς που θα ισχύσει Επίση, κάποια κρατημέλη θέλουν να βολέψουν τους δικούς τους ή τον εαυτό του τέλο πάντων και δεν θα πρέπει να υπάρξει μια ούτως πριν εναρμόνιση προς τα κάτω. Θα πρέπει επομένω να θωρακίσουμε την πρόταση της Κομισιόν και έτσι να κάνουμε αυτό που περιμένει ο κόσμος, δηλαδή να καταπολεμήσουμε την φοροδιαφυγή από τις εταιρείε παρά τις επιφυλάξεις. Εμείς θα επιψηφίσουμε την έκθεση και θέλουμε να υπάρξει ευρεία συνένεση και μεγάλη πλειοψηφία. Η αρχική πρόταση να είναι το ξεκάθαρο μήνυμα που θα στείλουμε για το θέμα μας στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κάποιο εκπρόσωπο της EFTD. Υπάρχει εκπρόσωπος του ENF. Θα ήθελε κάποιος να λάβει το λόγο εξ όμως της ομάδας αυτής. Όχι, εντάξει, επανέρχομαι στον εισηγητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, όπως καταλάβατε έχουμε τον ίδιο στόχο όλοι να αντιμετωπίσουμε τη φόρα αποφυγή. Οι μέθοδοι που προτείνονται για να γίνει κάτι τέτοιο βέβαια είναι πολύ διαφορετικές και δεν είναι δεδομένο το να τις ε, συγχωνεύσει κανείς σε μια συμβιβαστική λύση. Τώρα, για να διευκρινίσω κάτι, την Παρασκευή είχαν σταλεί οι συμβαστικέ τροπολογίε και ο κατάλογο ψηφοφορία. Αν υπάρχουν ακόμα Διαφωνίε και συζητήσει είναι γιατί προσπαθώ να βρω τη μεγαλύτερη <clears throat> δυνατή συμφωνία και με το ΕΛΚ που είναι η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι άλλε πολιτικέ ομάδε στο κοινοβούλιο μα δεν παίζουν ρόλο. Αυτό που είπε ο κύριο Τινίντε Μάιερ ισχύει για μένα. Θα γίνει αυτή η πολιτική συζήτηση απόψε το βράδυ. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε σε μια λύση. Αλλά δεν είναι μονάχα το θέμα του ποσοστού έκπτωσης για τα για το κόστος των επιτοκίων. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει εκ για μια συμβαστική λύση. Αλλά εγώ πιστεύω θα μπορέσουμε να βρούμε μια λύση για την ενώπιον της ε, αυριανής ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ λέει και ο Πρόεδρος. Ήταν μια σημαντική ανταλλαγή απόψεων και η ελπίδα μου είναι ότι επί της βάσης αυτής θα είναι δυνατόν να έχουμε μια ισχυρή θέση του Κοινοβουλίου αύριο, κύριε Νίντερμαϊερ. Θα χρειαστούν εδώ κάποιε διευκρινήσεις, λέει ο κύριο Νίτερ για το τι ακριβώς προτείνει ο εισηγητής. Αν υποστηρίξει τις συμβαστικέ λύσει όπως υπάρχουν αυτή τη στιγμή, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μπορέσει να εξασφαλίσει μια ισχυρή πλειοψηφία. Γιατί τουλάχιστον τρεις ομάδες εδώ, οι οποίες έχουν εκφραστεί σαφώς, δεν θα καλυφθούν από αυτές τις τροπολογίες. Επομένως μπορούν να γίνουν κάποιες ε, προσαρμογές στις συμβαστικές, αλλά κατά τα άλλα είναι επικίνδυνο να ψηφίσουμε αύριο. Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει να προτείνει λοιπόν ο σχετικά. Από ό,τι καταλαβαίνω, λέει ο πρόεδρος, η πρόταση του εισηγητή είναι ότι επί τη βάση των θέσεων που εκφράστηκαν εδώ στη συζήτηση τη σημαίνει, ιδίω από εσά, να επανέλθει και να προσπαθήσει να βρει κάποια λύση για την έκπτωση, για την εξυπηρέτηση δανείων, για τα επιτόκια. Έχουμε βέβαια ήδη τον κατάλογο ψηφοφορίας. Έχουμε προτάσεις για σύμβασικες τροπολογίες και είναι απόλυτα θεμητό να κάνουμε ψηφοφορία επί τη βάση αυτής της ε, θέσης. Δεν υπάρχει κάποιος Κανόνα του Κοινοβουλίου που λέει ότι πρέπει υποχρεωτικά να έχουμε μια ευρεία πλειοψηφία. Μπορούμε να ψηφίσουμε ούτω ή άλλω. Καταλαβαίνω ότι από πολιτική έποψη <clears throat> ο εισηγητή θα ήθελε να έχει μια ευρύτερη πλειοψηφία. Και αυτό θα το υποστήριζα και εγώ προσωπικά και νομίζω ότι οι πολιτικέ ομάδε πρέπει να προσπαθήσουμε να βρουν ένα κοινό έδαφο τουλάχιστον για κάποια σημεία τα οποία αναφέρθηκαν από τους εκπροσώπους των ομάδων. Μέχρι τώρα έχω ακούσει δύο πολιτικές ομάδες να είναι επικριτικά για τις συμβαστικές αυτές λύσεις. Δεν μπορώ εγώ να παρέμβω φυσικά στο σημείο αυτό. Είναι θετικό ότι έχουν γίνει κάποιες διευκρινήσεις για ορισμένα κρίσιμα σημεία και ότι είναι σημαντικό όλοι να ξέρουν ότι να εξακολουθήσει το Κοινοβούλιο να γίνεται αντιληπτό ως ένα θεσμικό όργανο το οποίο αγωνίζεται κατά της φοροαποφύγης. Είναι και πολιτικά και συμβολικά αυτό πολύ σημαντικό. Μπορώ να κλείσω λοιπόν τώρα τη συζήτηση. Καταλαβαίνουμε ότι οι πολιτικές ομάδες θα συναντηθούν μέσω των εκπροσώπων τους απόψε, οπότε θα υπάρχει δυνατότητα να εξετάσουν τον κατάλογο ψηφοφορία και προσβλέπουμε για στη συζήτηση των υπολείπων ανοιχτών σημείων μέσα <clears throat> από τους ε, σκιώδεις εισηγητές. Θα ήθελα λοιπόν να κλείσω αυτό το σημείο. Κύριε Λούκε, να έχετε το λόγο για διαδικαστικό θέμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω αγγλικά για να ευνοήσω την επικοινωνία. Αν κατάλαβα αυτά τα οποία λέγεται ο κ. Μπάτς προηγουμένως, υπήρξε απόφαση των συντονιστών να είναι έτοιμες μέχρι τις 3 η ώρα σήμερα οι συμβαστικές λύσεις. Υπάρχουν όμως συμβαστικέ λύσεις οι οποίες δεν έχουν ευρεία υποστήριξη Κάποιες ε, πολιτικές ομάδες λένε ότι τις δέχονται, άλλες ομάδες όχι. Εάν αυτές οι συμβαστικές λύσεις θα αλλάξουν σήμερα με συνομιλίες μεταξύ σοσιαλιστών και δημοκρατών, άλλες μικρότερες ομάδες μπορεί να μην εμπλέκονται σε αυτές τις ε, συμβαστικές λύσεις. Σήμερα λοιπόν που είναι 5 η ώρα σχεδόν δεν ξέρουμε τι θα ψηφίσουμε αύριο το πρωί. Αυτό είναι σαφής παραβίαση της συμφωνίας των συντονιστών. Σας ζητώ και πάλι λοιπόν η απόφαση να, να ληφθεί η απόφαση αναβολής της ψηφοφορίας και να μην γίνει αύριο ψηφοφορία, ώστε όλες οι ομάδες και όχι μόνο οι μικρές, οι μεγάλες ομάδες, να ξέρουν σε τι ψηφίζουν και να μπορούν να ψηφίζουν γνωρίζοντας περί τίνος πρόκειται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λούκε, αλλά σας ξαναλέω αυτό που σας είπα. Υπάρχει ένας κατάλογος ψηφοφοριών, υπάρχει ένας κατάλογος συμβιβαστικών λύσεων που έχει παρουσιαστεί, έλαβε χώρα μια συζήτηση και ο λόγος της συζήτησης είναι να δούμε αν χρειάζονται κάποιες προσαρμογές για να υπάρξει μια ευρεία πλειοψηφία. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν με ανοιχτό και διάφανο τρόπο και μπορεί αυτό να αφορά μονάχα μία ή δύο συμβαστικές λύσεις και μόνο. Θα δούμε λοιπόν τι θα προκύψει αύριο και η Επιτροπή μας έχει κάθε κυρίαρχο ρόλο Αξιολόγηση τη κατάσταση. Προς το παρόν όμω έχουμε μια ημέρησια διάταξη, έχουμε κάνει μια συζήτηση για τα θέματα αυτά. Το μόνο που μπορώ να κάνω λοιπόν είναι να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση και αύριο θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση αυτή και θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Αυτή είναι η απόφασή μου και γι' αυτό περνάμε στο επόμενο σημείο τη ημερησίας διάταξη. Λοιπόν, δημόσια ακρόαση για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων. Έχουμε μια πολύ σημαντική δημόσια ακρόαση, όπως ξέρετε, για το κέριο αυτό θέμα. Θέλω να χαιρετήσω όλους τους ομιλητές οι οποίοι δέχτηκαν την ε, πρόσκλησή μας και είναι έτοιμοι να συμβάλλουν στη συζήτηση αυτή. Αγαπητοί συνάδελφοι, αν θέλετε να μιλήσετε, σας παρακαλώ να φύγετε από την αίθουσα αυτή. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν όλους τους ε, ομιλητές οι οποίοι θα συμβάλλουν στη συζήτησή μας για αυτό το σημαντικό θέμα που είναι ένα σημαντικό συστατικό στοιχείο της Τραπεζικής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην εμβάθυνση της Νομισματικής και Οικονομικής Ένωσης και θα ήθελα να δώσω το λόγο, γιατί έχουμε καθυστερήσει λιγάκι, να δώσω το λόγο στον εισηγητή, στην εισηγήτρια την κυρία Εστέρ Ντελάγκε. Ευχαριστώ. Όπως ξέρετε έχω αρκετά πράγματα να πω για αυτό το θέμα. Τώρα δεν υπάρχει ώρα για εισαγωγή. Έχουμε καθυστερήσει ήδη και δεν θέλω να φάω άλλο χρόνο από τους ομιλητές μας. Προτείνω λοιπόν να ξεκινήσουμε με την ακρόαση, η οποία όπως ξέρετε αποτελείται από δύο μέρη πρώτα απ' όλα. Τι μορφή θα έπρεπε να έχει ένα ιδεώδες τέτοιο σύστημα και εξίσου σημαντικό, αν μπορούμε να συμφωνήσουμε στο πρώτο αυτό, πώς θα καταλήξουμε στη μορφή που θέλουμε. Και με την κατάσταση που έχουμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που δυστυχώς χαρακτηρίζεται από χαμηλή εμπιστοσύνη Θα μείνω λοιπόν σε αυτά για να ακούσουμε τους ε, ομιλητές μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και εγώ. Περνάμε λοιπόν απευθείας στην πρώτη συνεδρία πώς θα λειτουργήσει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Αγγίσης Καταθεσιών στην τελική του φάση. Καλή ερώτηση, δύσκολη. Δεν κουπέ Πρώτος ομιλητής, ε, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Εγγύησης Καταθέσεων, έχει τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Γκουαλχέρη. Χαίρομαι που είμαι εδώ, που με προσκαλέσατε στην ακρόαση αυτή. Να κάνω πρώτα μια εισαγωγή για το FD. Πρόκειται για μια αστική εταιρεία που συστάθηκε στο Βέλγιο το 2002 εκπροσωπούμε ε, όλα τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων στην Ευρώπη όλων των κρατών μελών της Ένωσης ε, και των χωρών ΕΟΧ, Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, οπότε όλες οι χώρες ε, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Συνεισφέρουμε λοιπόν στην σταθερότητα του συστήματος και συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Για τα ζητήματα αυτά βεβαίως ε, δεν έχουμε ακόμα καταλήξει το πώς θα λειτουργήσει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Αγγίζης Καταθέσεων στην τελική του μορφή, γιατί είναι καινούριο το ζήτημα. Θα ήθελα απλά να εκφράσω κάποιες απόψεις ε, σήμερα και θα αφαιρθώ κυρίως βεβαίως στην δική μας Έχω επίσης καταθέσει στα πρακτικά το επίσημο έγγραφό μας ε, για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων, οπότε υπάρχει αναλυτικά η απόψή μας. Προσωπικά ε, θα ήθελα να μιλήσω στο πάνελ 2 γιατί θα ήταν πιο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα φτάσουμε στο ΙΔΙΣ και ποια θα είναι η τελική του μορφή, γιατί δεν έχω πιστεί ότι θα φτάσουμε ως εκεί και τι μορφή θα έχει και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Αλλά αφού εδώ με προσκαλέσατε στο πρώτο πάνελ θα μιλήσω για αυτά τα οποία μου ζητήσατε. Εμείς έχουμε πολύ συγκεκριμένες ε, θέσεις, οι οποίες συμφωνούν ε, όλα μας τα μέλη για το ότι δηλαδή η Κομισιόν θα έπρεπε να κάνει μια αξιολόγηση αντικτύπου, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει. Να σας πω λοιπόν κάποια πράγματα από τη σχετική μας δήλωση. Ανεξαρτήτως της μορφής και της αναγκαιότητας που θα λάβει το σύστημα αυτό, τα μέλη μας θεωρούν πως η αξιολόγηση αντικτύπου του 2010 της Κομισιόν δεν αποτελεί επαρκή βάση για την πρόταση της Κομισιόν καθώς πλέον έχει τεθεί σε ισχύ το Ευρωπαϊκό, ο Ευρωπαϊκός Σταθερότητας και το GSST και έχει αλλάξει ουσιαστικά το νομικό πλαίσιο από το 2010 άρα θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση αντικτύπου και μια ανάλυση κόστους ωφέλους. Αυτή είναι λοιπόν η άποψή μας εδώ πέρα ότι δεν έχει γίνει η σωστή αξιολόγηση αντικτύπου και η κατάλληλη διαβούλευση και θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει. Και θεωρούμε πως ε, δεν μπορεί ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να υποκαταστήσουν αυτές τις εργασίες πρέπει να κάνει η Κομισιόν γιατί η Ολλανδική Προεδρία έχει θέσει 18 τεχνικά ερωτήματα της Κομισιόν και από όσο αντιλαμβάνομαι η Κομισιόν έχει απαντήσει μόλις σε ένα μέχρι στιγμής. Η ρευστότητα επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική. Η Κομισιόν έχει αναφερθεί σε πιθανά μεγάλα τοπικά σοκ, κάτι το οποίο σημαίνει πως ίσως να μην υπάρχει επαρκής οικονομική στήριξη από τα κράτη-μέλη ή και από οποιοδήποτε άλλο θεσμικό όργανο. Επίσης, θεωρούμε πως η ρευστότητα είναι βασικός παράγων, αλλά βεβαίως ε, δεν μιλάμε μόνο για ρευστότητα, μιλάμε και για το πώς θα μοιραστούμε τις ζημιές και αν χρειαζόμαστε έναν τέτοιο μηχανισμό στο μέλλον. Κατά την άποψή μας, με την ε, εισαγωγή της ε, προτίμησης των κατατεθών υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυνατότητα να πιθανότατα συγχωρείτε, τα συστήματα ασφάλισης ε, καταθέσεων να ανακτήσουν ε, τελικά το 100% των ε, συνεισφορών τους. Οπότε δεν μιλάμε για ζημίες, αλλά ουσιαστικά για ρευστότητα η οποία θα απαιτηθεί. Οπότε, μήπως επαρκεί ο δανεισμός αντί για ένα μηχανισμό ο οποίος θα μοιράζει τις ζημιές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ πέρα το ότι οι διαδικασίε χρεοκοπία ε, στα κράτη-μέλη θα πρέπει να εναρμονιστούν, να υπάρξει ανάκτηση των στοιχείων ε, του ενεργητικού των εταιριών στι διαδικασίε χρεοκοπία, γρηγορότερα σε όλα τα κράτη-μέλη. Επίση, η χρηματοδότηση. Πολύ σημαντική πτυχή. Ο προτινόμενο μηχανισμό μειώνει το κίνητρο να πάει κάποιο πέρα από το 0,8%. Γιατί να το κάνει κάποιο εάν τα άλλα κράτη-μέλη θα μείνουν στο 0,8%. Πολύ σημαντικό αυτό. Το παρατηνόμενο σύστημα επίσης ε, αγνοεί τις δεσμεύσεις ε, πληρωμών ε, που έχει εδώ πέρα εισαγάγει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και εφαρμόζουν τα κρατημέλη. Δεν γνωρίζει τέτοιε δεσμεύσει πληρωμών και πρόκειται για στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ των ασφαλιστών καταθέσεων εντός και εκτός Ευρωζώνης που οι δεύτεροι μπορούν να να εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τέτοιε δεσμεύσει. Είμαστε λοιπόν υπέρ ε, των συνεισφορών οι οποίες ε, θα βασίζονται στην στάθμιση του κινδύνου, αλλά θα πρέπει βεβαίως ε, να μιλάμε για το επίπεδο 1. Και βεβαίως δεν είναι στην πράξη δυνατή η διπλή εισφορά θα μπορούσε θεωρητικά να μεταφερθούν οι εισφορές αυτές από το εθνικό επίπεδο στο ευρωπαϊκό σύστημα, αλλά μετά μπαίνουμε σε πολύ περίπλοκα ζητήματα και υπάρχουν συντάγματα κρατών μελών που δεν επιτρέπουν λεφτά τα οποία έχουν συλλεγεί για ένα συγκεκριμένο σκοπό να μεταφερθούν στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, κάποιες προσωπικές απόψεις για την πρόταση για το ευρωπαϊκό σύστημα. Η νομική βάση αμφισβητείται. Υπάρχει έντονη συζήτηση και ένας άλλος ειδικό που βρίσκεται εδώ πέρα έχει δημοσιεύσει μια εργασία για την νομική αυτή βάση η οποία αμφισβητεί όπως είπαμε την νομική βάση θα προτιμούσα να έχουμε μια στιβαρή νομική βάση για την πρόταση αυτή η μείωση του κινδύνου θα πρέπει πρώτα να αντιμετωπίσει τα ιστορικά ζητήματα που υπάρχουν ακόμα επίσης το έντις στρεβλώνει τον ανταγωνισμό μεταξύ αυτών που είναι εντό και εκτό. δηλαδη δηλαδή κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία δεν θα ανήκουν στο σύστημα θα χρησιμοποιούν δεσμεύσει πληρωμών ενώ τα μέλη τη Ευρωζώνης δεν θα μπορούν πλέον. Η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαλέξει δηλαδή μεταξύ του στόχου 0,8%, 0,5% ή και 0,0% όπως το Ηνωμένο Βασίλειο. Εν τω μεταξύ, τα μέλη της Ευρωζώνης πρέπει να μείνουν στο 0,8% χωρίς ε, δεσμεύσεις Ένα Εναλλακτικά μέτρα, ένα βασικό σημείο για τους ασφαλιστές ε, καταθέσεων και ε, να σας υπενθυμίσω εδώ πέρα πως το Κοινοβούλιο έβαλε ακριβώς αυτό το θέμα στην πρόταση του GDST. Δεν ήταν αυτό στην πρόταση της Κομισιόν του 2010. Το Κοινοβούλιο τα εισήγαγε και δεν θα υπάρχει πλέον αυτή η δυνατότητα στο μέλλον. Μόνο εάν χρηματοδοτηθούν από επιπρόσθετα κονδύλια τα οποία θα πρέπει να, τα... να είναι πάνω από το 0,8%. Εν τω μεταξύ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει τη δυνατότητα να συλλέγει 0,8, 0,5 ή 0,0 και να χρηματοδοτήσει έτσι εναλλακτικά μέτρα. Οι μηχανισμοί ασφάλισης ε, καταθέσεων θα πρέπει να παίξουν έναν πιο ενεργητικό ρόλο στο Ναι, έχουν τελειώσει τα πέντε λεπτά. Πώς θα λειτουργήσει λοιπόν στην τελική του σταθερή φάση το σύστημα αυτό. Πρόκειται λοιπόν για ένα σύστημα το οποίο βράχει πρόθεσμα, ε, μέσω πρόθεσμα θα μπορέσει να λειτουργήσει σε αμοιβαίο δανεισμό. Μακροπρόθεσμα θα πρέπει να αναφερθούμε στο άρθρο 19.5 της ε, σχετικής οδηγίας η οποία βεβαίως ε, μιλάει για ένα σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο της Ευρωζώνης. Και βεβαίως εάν ο αμοιβαίος δανεισμός ε, δεν αποδειχθεί επαρκής τότε θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για κοινό κίνδυνο, κοινή ανάληψη κινδύνου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα ο δεύτερος σωμητής είναι ο κύριος ε, Βόλ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα να είμαι εδώ και να μπορέσω να αναφερθώ στη μακροχρόνια σχεδίαση του ΙΝΤΙΣ, του συστήματος ε, γίνησης καταθέσεων, παρά το γεγονό ότι καταλαβαίνω για την Κομισιόν ορίζοντας είναι πολύ μακρινός, 2024-2025 υπάρχουν πολλά εμπόδια που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και πρέπει να σκεφτούμε και για όλα αυτά τα θέματα. Θα κάνω μερικέ γενικέ παρατηρήσει για την εγγύηση, των, κατά την ασφάλεια των κατηθέσεων και γιατί χρειαζόμαστε ένα τέτοιο σύστημα. Πρώτα απ' όλα, ποιο είναι ο ρόλο τη εγγύηση των καταθέσεων για μένα. Είναι πολύ σημαντικό το να καταλάβουμε ότι αυτό είναι κυρίως ένα εργαλείο για να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη των καταθετών στις τράπεζες και στην σταθερότητα των τραπεζών αυτών. Φυσικά είναι κύρια ευθύνη των τραπεζών να εξασφαλίσουν αυτή την εμπιστοσύνη. Σε ορισμένε περιπτώσει όμω δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Δεν μπορούν από μόνε του να το εξασφαλίσουν. Εκεί χρειαζόμαστε ένα σύστημα εγγύηση καταθέσεων. Το δεύτερο ερώτημα είναι να χρειαζόμαστε ένα τέτοιο ευρωπαϊκό σύστημα για την εγγύηση των καταθέσεων. Για μένα υπάρχουν τρία επιχειρήματα που συνοδορούν υπέρ ενό ευρωπαϊκού συστήματο. Καταρχήν το θέμα του μεγέθου. Η τα σύστημα ασφαλίσεις δουλεύουν καλύτερα όσο μεγαλύτερη κάλυψη έχουν. Αυτό είναι ο νόμος των μεγάλων αριθμών, αν θέλετε. Αν έχετε μονάχα εγγύηση για δύο ή τρεις τραπέζες, τράπεζες και μία από αυτές επηρεάζεται από κάποιο πρόβλημα, είναι πολύ δύσκολο να χρηματοδοτηθεί η εγγύηση και να ανανεωθούν τα κονδύλια τα οποία χρειάζονται. Θέλετε να έχετε ένα μεγάλο δείγμα τραπεζών και αυτό επομένως ευνοεί ένα ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης καταδέσεων. Το δεύτερο είναι το θέμα της συνεκτικότητας. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα σύστημα όπου η εποπτεία των τραπεζών είναι κεντρική με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ενώ η ασφάλεια των καταθέσεων είναι αποκεντρωμένη στα κράτη-μέλη. Γιατί αυτό σημαίνει ότι σε τελική ανάλυση μια απώλεια εποπτείας, μια αστοχή εποπτείας σε κεντρικό επίπεδο μπορεί να οδηγήσει στην ανάγκη και φορολογούμενοι να πληρώσουμε τα σπασμένα για μια λανθασμένη απόφαση που γίνεται στη Φραγκφούρτη. Τρίτο στοιχείο, η αποσύνδεση των τραπεζών από το κρατικό χρέος. Αυτό είναι και ένας από τους βασικούς στόχους της τραπεζικής έννοιας και αυτό αναφέρεται σε επίσημες και σε ανεπίσημες δηλώσεις ότι ο στόχος είναι να αποσυνδεθούν οι τράπεζες από τα κρατικά ομόλογα και επειδή η εμπιστοσύνη που έχετε σε ένα σύστημα εγγύησης καταθέσεων εξαρτάται και από, την, από το κράτος το οποίο εφαρμόζει αυτήν την εγγύηση, δεν είναι εύκολο χωρίς ένα ευρωπαϊκό σύστημα να υπάρξει πλήρης αποσύνδεση. Ένα τελευταίο σημείο είναι η διαχείριση των κρίσεων. Ξέρουμε ότι η συνθήκη του ESM προβλέπει ότι αν υπάρξει αφαιρεγγιότητα μιας κυβέρνησης δεν μπορεί να υπάρξει ε, χρηματοδότηση εάν δεν υπάρξει προηγουμένως συμμετοχή των καταθετών και των ομολογιούχων του κρατικού χρέους. Αυτό κάνει πιο εύκολη κάπως την ε, επίλυση των κρίσεων. Θέλω να αναφέρω εδώ και το θέμα των ε, κρατικών ομολόγων που βρίσκονται στα χέρια των τραπεζών. Είναι κάτι το οποίο έχει τύχει μεγάλη ε, προσοχή στη συζήτηση, αλλά είναι ένα πάρα πολύ Πολυδέταλο θέμα. Ξέρουμε ότι το κρατικό χρέος συνήθως κρατιέται από τις τράπεζες της ίδιας χώρας η οποία εκδίδει αυτό το χρέος. Το πρόβλημα είναι ότι εάν δεν μειώσετε την έκθεση των τραπεζών αυτών στο εθνικό κρατικό χρέος και συγχρόνως έχετε ένα ευρωπαϊκό σύστημα υγιής καταθέσεων, ο κίνδυνος μπορεί να είναι να υπάρχει αυτό το σύστημα ασφάλισης το οποίο θα πρέπει να καλύψει προβλήματα τα οποία προκύπτουν από την εθνική φορολογική ή δημοσιονομική πολιτική πάνω στην οποία δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να ασκηθεί πίεση. Επομένως, με τον τρόπο αυτό θα καλύπτονται απώλειες οι οποίες προκύπτουν από την πολιτική των κρατών μελών. Γι' αυτό η δημιουργία ενός καθαρά, ενός πλήρως ευρωπαϊκού συστήματος ε, ασφάλειας καταθέσεων απαιτεί και μια σημαντική μείωση της έκθεσης των τραπεζών στο κρατικό χρέος της χώρας τους. Τώρα υπάρχει συζήτηση αν θέλουμε μια πλήρη, ε, ένα πλήρες σύστημα ασφάλισης ή αντασφάλισης. Ένα σύστημα αντασφάλισης μπορεί μόνο σε κάποιο περιορισμένο βαθμό να αποσυνδέσει τις τράπεζες από το κρατικό χρέος, αλλά δεν μπορεί να καλύψει απόλυτα αυτή την αποσύνδεση. Θα έλεγα όμως ότι υπάρχει λογική θα να ξεκινήσουμε με ένα σύστημα αντασφάλισης, γιατί είναι πολλές χώρες οι οποίες έχουν ιδιαιτερότητε στα εθνικά συστήματα και δίνουν και ειδικέ μεταχειρήσεις σε ό,τι αφορά την προστασία των καταθέσεων και το αναφέρατε προηγουμένως. Και έχουμε επίσης και μια πραγματική κατακαιρμάτιση των συστημάτων ασφάλισης ε, καταθέσεων, οπότε το σύστημα της αντασφάλισης μπορεί να είναι μια καλή αφετηρία επειδή δεν έχω χρόνο, να αναφερθώ σε ορισμένα ενοιολογικά στοιχεία για τους κανόνες του Μπέιλιν, της συμμετοχής των καταθετών και ομολόγου ιούχων. Ένα επιχείρημα κατά του ευρωπαϊκού συστήματος ε, καταθέσεων υπάρχει μια ιεραρχία των ε, αυτών οι οποίοι πρέπει να συμβάλλουν. Λένε ορισμένοι ότι δεν πρέπει να υπάρχει ασφάλεια στις καταθέσεις, αλλά αυτή η διαδικασία ασφάλειας των καταθέσεων έχει σαν στόχο να δημιουργήσει εμπιστοσύνη. Κανείς δεν ξέρει πλήρω το χαρτοφυλάκιο μιας τράπεζας και δεν ξέρει ποιος θα είναι αυτός ο οποίος έχει λιγότερο εξασφαλισμένο χρέος και επομένως θα πρέπει να πληρώσει πριν από αυτόν τον ίδιο. Επομένως το θέμα της ασφάλειας έχει σαν στόχο να αυξήσει την εμπιστοσύνη των καταθετών. Το πρώτο τελευταίο μου λοιπόν σημείο είναι σε σχέση με τη σημασία του να υπάρχει μια ε, στερεή, στερεά ε, βάση σε νομικό και πολιτικό επίπεδο. Εδώ το πιο σημαντικό είναι ότι αν θέλουμε να έχουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης καταθέσεων πρέπει να βασίζεται σε μια ισχυρή πολιτική και νομική βάση, γιατί αν είναι αδύναμη αυτή η βάση του, δεν θα αποκομίσει την εμπιστοσύνη των καταδετών. Ή κρατάμε το εθνικό σύστημα ή έχουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα. Άμα έχουμε μια μεσοβέζικη λύση η οποία δεν είναι και τεχνικά αξιο... αξιόπιστη, δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα. Εν κατακλείδη λοιπόν θα έλεγα ναι, είναι απαραίτητο, είναι θετικό να έχουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα κατα... εγγύησης καταθέσεων, αλλά μονάχα εάν γίνει αυτό με σωστό τρόπο και εάν υπάρχει μια μεσοβεζικη λυση η οποια δεν ειναι και τεχνικα αξιοπιστη δεν μπορουμε να πετυχουμε τιποτα εν κατακλειδη λοιπον θα ελεγα ναι ειναι απαραιτητο ειναι θετικο να εχουμε ενα ευρωπαικο συστημα κατα βάση για αυτό το σύστημα και αν εξασφαλιστεί ότι με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και θα αντιμετωπιστεί το θέμα σύνδεση των τραπεζών με το κρατικό χρέο. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Ευχαριστούμε τον Ντάνιελ Γκρόζο για τη Σκητάλη που είναι διευθυντή από το Κέντρο Μελετών Ευρωπαϊκή Πολιτική. Σα ευχαριστώ πολύ. Χαρά βρίσκομαι εδώ και να συνεχίσουμε τώρα ε, αυτήν την άνηση προσέγγιση του πάνελ, Άνηση, τέλο πάντων πλευρά ε, εθνική προέλευση. Ακριβώς, ε, όπω είπε ο, ο Γκίντερ, θα πρέπει να δούμε τώρα το πόσο επιθυμητό, ευκταίο είναι να έχουμε ένα τέτοιο σύστημα ασφάλιση καταθέσεων. Διότι το πρόβλημα, όπως καλά γνωρίζουμε, είναι το εξής. Ότι όταν έρθει η με στιγμή, όταν δηλαδή ε, σοβεί μια μεγάλη κρίση, τότε οι κυβερνήσεις πελαγώνουν ακριβώ την ώρα που χρειάζεται να επιστρατεύσουν ό,τι εργαλεία έχουν ούτω ώστε να επαναφέρονται σταθερότητα στο τραπεζικό. Βεβαίω, και κάτι χρειάζεται. Βέβαια, το θέμα της αντασφάλιση ή αυτασφάλιση είναι πάρα πολύ σημαντικό και όχι μόνο σαν μεταβατικό ε, μέτρο, αλλά και σαν μια πάγια λύση. Κατά τη γνώμη μου αυτή η προσέγγιση με την αντασφάλιση επίσης καλύπτει και το θέμα της επικουρικότητας διότι τα προβλήματα αυτά τα οποία έχουμε με την ασφάλιση των καταθέσεων είτε αφορούν πολλές μικρές τράπεζες ή, μεγαλύτερα, ευρύτερα προβλήματα με ή μεγαλύτερες τράπεζες και έχουν συστημική μόρφη. Άρα έχουμε πάρα πολλές μικρές ε, τράπεζες που φυσικά είναι περισσότερες αλλά αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί σε εθνικό επίπεδο και από την άλλη μεριά έχουμε τα επιμέρου συστήματα ασφαλής των καταθέσεων που υπάρχουν πολλές φορές κάποιες χώρες έχουν περισσότερα από ένα σύστημα. Επομένως υπάρχουν ε, καλύψεις από πολλές πλευρές, ε, λειτουργούν έβρα. Όμως, όταν έχουμε το άλλο πρόβλημα δηλαδή, όταν έχουμε συστημικό πρόβλημα σε εθνικό επίπεδο, ε, τότε θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός και να εξασφαλίζει ότι το Εθνικό Σύστημα Ασφάλισης Εγγυήσεων θα μπορεί να είναι αξιόχρονο, θα μπορεί να διασώσει, να εξασφαλίσει. Αυτό πάνε να πει αντασφάλιση και αυτασφάλιση. Ότι δηλαδή ο αντασφαλιστής σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα παρεμβαίνει μόνο εάν έχουμε ένα μείζον πρόβλημα. Ακριβώς όταν το εθνικό σύστημα έχει φτάσει στα ωριά του. Άρα, αυτή η αντασφάλιση θα πρέπει να ενταχθεί στην γενικότερη προβληματική να ασφαλιζόμαστε όσον αφορά τις μείζονες διαταράξεις των κρατών μελών. Να και ποιο είναι το πρόβλημα στην Ευρωζώνη. Αλλά και μέχρι ένα σημείο στη όλη Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή ότι στη φυσιολογική ροή των πραγμάτων τα κράτη-μέλη μπορούν να αντιμετωπίσουν τις κυκλικές ε, διαταράξεις. Ε, με αυτά για όταν όμως τα πράγματα χειροτερεύουν, όταν υπάρχει αποκοπή από τις χρηματαγορές, ε, τότε χρειάζεται η στήριξη και η διάσωση. Να, τι θα μπορούσε να γίνει με αυτή την προσέγγιση της αντασφάλισης και οπότε δεν χρειάζεται κάποια περίπλοκη δομή για αυτήν την ασφάλιση και αντασφάλιση διότι ο σκοπός του ασφαλιστή θα είναι να ασκεί κάποιο είδου εποπτικό ποιοτικό έλεγχο όσον αφορά τους εθνικούς μηχανισμούς διάσωσης. Κάτι ε, το οποίο ισχύει και σε επίπεδο εμπορίου. Το θέμα δεν είναι επομένως έναντι ποιου κινδύνου ασφαλίζει κανείς, αλλά θα πρέπει κανείς να δει πώς γίνεται η διαχείριση του κινδύνου. Ποιο είναι το επιχειρηματικό μοντέλο των ε, ε, ασφαλιζομένων που καλύπτει ο ασφαλιστής. Άρα, ο αντασφαλιστής θα πρέπει ακριβώς να αναλύσει την δομή του τραπεζικού συστήματος στην χώρα που κάθε φορά ε, πρέπει να καλύψει. Θα πρέπει να δει πόσο στέρεο είναι το σύστημα, φυσικά και τι επιδόσεις έχει το κράτος για να είναι ο δανειστής τελευταίας καταφυγής, τελευταία λύση και από του ασφαλιστή θα πρέπει να εξεταστούν όλες οι λεπτομέρειες. Ό,τι νομοθετικά ισχύει. Στο πτωχευτικό δίκαιο ας πούμε, το εθνικό, ό,τι τέλος πάντων επηρεάζει το πού θα καταλήξει μια ε, προβληματική κατάσταση κάποιας τράπεζας. Οπότε η, ασφάλιση ε, βέβαια των καταθέσεων είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την ανακεφαλαιοποίηση γιατί στη θεωρία εάν έχουμε κάποια ανακεφαλαιοποίηση σε κάποια τράπεζα ε, τότε ενεργούμε με επένδυση που θεωρητικά θα αποδώσει ε, θα αποδώσει και εγώ και έχουμε και τον και το Συμβούλιο Σαρμπή και λοιπά. Τώρα όμως ε, στην ασφάλιση ε, ελαχιστούμε τον κίνδυνο, τον φρενάρουμε, αλλά υπάρχει ζημία. Και άρα στην ασφάλιση καταθέσουμε θέλουμε ένα σύστημα το οποίο στο εθνικό επίπεδο διατηρεί τα πράγματα υπό έλεγχο και οπότε υπάρχει ετοιμότητα παρέμβαση όποτε έχουμε ε, κάποια μίζωνα κρίση που χτυπάει τη χώρα σαν να υπάρχει μια ασφάλιση ε, οπότε για τις μικρές κρίσεις ε, κάποιος, ε, ε, υπάρχει όριο δηλαδή στην ασφαλιστική σύμβαση και καλύπτεις μόνο στις μικρές ζημιές για τις μεγάλες ζημιές παρεμβαίνει ο ασφαλιστής. Άρα θα πρέπει να γίνει η, η ελάχιστη των παρεμβάσεων σε εθνικό επίπεδο και έτσι να έχουμε ένα σύστημα που να καλύπτει την συστημική σταθερότητα αυτό ακριβώ που προαναφέρθηκε. Βέβαια τα μεσοβούνα χρόνια θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την υπερβολική συγκέντρωση του ρίσκου που παίρνουν οι τράπεζες ε, ως προς το κρατικό χρέος και άρα θίγεται το ισολογισμός τους. Επομένως, δεν νομίζω ότι αν τα ασφάλισε και από τα ασφάλισε θα πρέπει να θεωρηθεί μια πάγια λύση. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε και τώρα για μεγάλη μας χαρά να δώσουμε στον κύριο το λόγο που προέρχεται από το Συμβούλιο Εξυγένσης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τι μορφή θα έχει το σύστημα εγγύησης καταθέσεων στην τελική του μορφή. Πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, οπότε θα ξεπεράσω την ερώτηση για τη μείωση του ρίσκου και βεβαίως μιλώντας για το ενιαίο Συμβούλιο Διάσωσης βεβαίως είμαστε υπέρ και ακούστηκαν κάποια επιχειρήματα αλλά θα προσπεράσω αυτή την συζήτηση και θα ξεκινήσω με κάτι το θετικό αυτή τη στιγμή στα περισσότερα κράτη-μέλη έχουμε μεταφέρει την ε, οδηγία για την εγγύηση των καταθέσεων στο εθνικό δίκαιο. 12 μήνες μόλις μετά την προθεσμιακά, το οποίο είναι επίτευγμα. Οπότε έχουμε μια αφετηρία, έχουμε μια σοβαρή βάση για τα επόμενα βήματα. Την πρόταση της Κομισιόν την ξέρουμε και χωρίς να την επαναλάβω θα ήθελα να δούμε τα πράγματα κάπως ευρύτερα και εδώ να διαφωνήσω λίγο κάπως με κάτι το οποίο είπε ένας θα ήθελα να θυμόμαστε πως αυτά τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε μακροπρόθεσμα είναι κάπως ευρύτερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μέσω του BRD οικοδομήσει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο διάσωσης αλλά είναι μόνο ένα κομμάτι του συστήματος και βεβαίως ε, δεν θέλουμε ποτέ να έχουμε αποδόσεις από την επένδυση αυτή. Αλλά είναι ένα καθεστώς ε, για μεγαλύτερες τράπεζες οι οποίες έχουν κρίσιμες λειτουργίες και πιθανώς συστημικές επιπτώσεις. Τούτων λεχθέντων πρέπει να υπάρχει μια οικονομική απάντηση για τις μικρότερες τράπεζες και το σύστημα εγγυήσεων καταθέσεων είναι κατά βάση ένα σύστημα εμπιστοσύνης, το θεμέλιο για τις μικρότερες τράπεζες να ε, έχουν ε, θα έλεγα ίσους όρους οπότε ε, θα μιλούσαμε για ένα τρίγωνο χρειάζεται δηλαδή το σύστημα των ίσεων καταθέσεων και ένα αποτελεσματικό σύστημα διάσωσης για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα δύο προηγούμενα. Οπότε, όπως είπα, όταν μιλάμε για μια σταθερή φάση, υπάρχουν τρεις πτυχές, τρία μέρη του τριγών. Σχεδιάζοντας λοιπόν το Ευρωπαϊκό Αυτοσύστημα Εγγύησης Καταθέσεων πρέπει να φροντίσουμε οι τράπεζες οι οποίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να πάνε στην ε, διάσωση, δηλαδή οι μικρότερες τράπεζες θα μπορούν να μπουν στην διαδικασία χρεοκοπία και έτσι θα μπορέσουν τα συστήματα εγγύηση καταθέσεων ε, να παρέχουν ε, μια συνέχεια για τους καταθέτες. Οπότε θα πρέπει να δούμε το τι προβλέπει το άρθρο 11.6 της ε, οδηγίας, τα εναλλακτικά μέτρα και να εφαρμοστούν αυτά, αν πάμε για ένα ευρωπαϊκό σύστημα, στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Για να υπάρχει, όπως σας είπα, μια συνέχεια των υπηρεσιών και όχι απλά να πληρώνουμε. Εδώ πρέπει λοιπόν να το σκεφτούμε πολύ περισσότερο το θέμα και για να μείνω εντός των πέντε λεπτών το επόμενο θέμα είναι όταν κοιτάμε το ποιος πρέπει να κάνει τι. Η πρόταση της Κομισιόν προτείνει να δοθεί η διοίκηση στο Συμβούλιο Συστημικής Σταθερότητας ακολουθώντας το Αμερικανικό σύστημα μπορούμε να έχουμε διάφορα βήματα, μπορεί να προηγηθεί η αντασφάλιση ή να παγώσει, αλλά βεβαίως αυτός ο οποίος θα κάνει την αντασφάλιση δεν κοιτάει λίγο το επιχειρηματικό μοντέλο και πληρώνει, πληρώνει μόνο για θεμητά αιτήματα, παραδείγματος χάρη στην περίπτωση στην οποία υπάρχει δόλος ε, δεν ε, καλύπτει ποτέ. Οπότε εδώ πέρα θεωρώ πως θα πρέπει να συνδυαστούν ε, τα δύο αυτά για να υπάρχει μια δυνατότητα διάσωσης και για τις μικρότερες και για, και για τα μεγαλύτερα πιστωτικά ιδρύματα και από την άλλη θα έλεγα πως ε, εξπακούεται στην πλευρά της διάσωσης πως υπάρχει σοβαρός ρόλος για τα εθνικά συστήματα εγγύησης καταθέσεων που θα πρέπει να συνεχίσουν να τον παίζουν γιατί βεβαίω είναι δρεωμένα όλα αυτά στο εθνικό δίκαιο και τελευταίο υπάρχει και το θέμα της χρηματοδότησης αυτών των συστημάτων γιατί από εκεί προκύπτει βεβαίως και η εμπιστοσύνη όταν υπάρχει χρηματοδότηση, όχι όταν είμαστε στην ιδέα. Θα σταματήσω εδώ λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Βλέπω ότι υπάρχει και σημαντική σύγκληση σε ό,τι αφορά τα προτινόμενα εναλλακτικά μέτρα. Αυτό είναι σημαντικό. Μπορούμε να επανέλθουμε τώρα στην εισηγήτρια και τους σκιώδες. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Έστερ Ντελάγκε. Για να επανέλθω στο τελευταίο σημείο <clears throat> για το σημαντικό ρόλο που επέχουν τα εθνικά συστήματα εγγύησης καταθέσεων και το πώς χρηματοδοτούνται και πώς λειτουργούν. Επανέρχομαι σε αυτό το τελικό λοιπόν σχόλιο. Ίσως ο κύριος Κουπάη θα μπορούσε να πει κάτι γι' αυτό γιατί αυτός έχει τη γενική εικόνα των εθνικών συστημάτων. Πώς μπορεί λοιπόν <clears throat> να εκτιμήσει τη γενική κατάσταση σε ό,τι αφορά την ε, ε, μεταφορά της ε, διεθνούς ή ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Δεν μας είπε όμως πως βλέπει την πραγματική λειτουργία και χρηματοδότηση των εθνικών συστημάτων, όχι να μας πει για όλες τις χώρες προφανώς, αλλά πώς βλέπετε να υπάρχουν διαφορές μεταξύ διαφορετικών ομάδων χωρών σε ό,τι αφορά την προσέγγιση που ακολουθούν. Στον κύριο Βόλφ σε αυτό που είπε για αυτούς που είναι μέσα και <coughs> έναντι αυτό που είναι έξω από την ε, Τραπεζική Ένωση. Το έχετε παρουσιάσει το θέμα αυτό και στην Επιτροπή μας σε άλλες περιπτώσεις, αλλά πώς βλέπετε αυτή την πρόταση για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων που ουσιαστικά αφορά τις 19 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι μέσα στο ευρώ και όχι τις 28. Μπορείτε να δώσετε εδώ κάποια σχόλια. Και για τον κύριο Γκρός αν θα μπορούσε να συγκρίνει αυτά που είπε για το σύστημα αντασφάλισης με αυτά που είπε ο κ. Κούπερ για, την, ε, για τον κατά κάποιο τρόπο επιμερισμό της ασφάλισης μεταξύ των κρατών μάλλον. Κυρία Κιόνιχ, επίσης, συνήθως στην Επιτροπή μας μιλάτε για και κάποια άλλα θέματα. Ίσως θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε γιατί θα ήταν σημαντικό να διατηρήσουμε ένα ελάχιστο επίπεδο 8% για το κεφάλαιο το οποίο μπορεί να υποβληθεί σε Μπέιλιν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. και για τις εθνικές επιλογές και διακριτική ευχέρεια. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να κάνετε κάποια σχόλια για αυτά. Θα πρέπει να παραμείνει κάποιο περιθώριο εσείς λέτε ότι πρέπει να υπάρχει λιγότερο περιθώριο για εθνική διακριτική ευχέρεια. Πώς ακριβώς το βλέπετε αυτό, μέχρι πού θα πρέπει να προχωρήσουμε προσπαθώντας να έχουμε ή δυνατόν κοινού κανόνες για τα θέματα αυτά. Θα είχα πολύ περισσότερες ερωτήσεις να κάνω βέβαια, <clears throat> κύριε Πρόεδρε, αλλά προς το παρόν σταματώ εδώ και απλώς να ευχαριστήσω τους ομιλητές για τη συμβολή τους. Η Ελίζα Φερέιρα έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ και όλους τους ομιλητές. Ξεκινώ με τον κύριο Κούπε. Και συνεχίζω στο ερώτημα που έθεσε η κυρία Ντελάγκε. Όταν βλέπετε διαφορετικά συστήματα, πώς τα συγκρίνετε σε επίπεδο λειτουργίας και σε επίπεδο διαφάνειας. Πώς εξασφαλίζετε <clears throat> ότι υπάρχει ένας ισότιμος ανταγωνισμός. Υπάρχουν διαφορές, θα πρέπει να τις λάβετε υπόψη ή όχι για τον κύριο Βόλφ. Σας ευχαριστώ για το γεγονός που μας υπενθυμίσατε τα διαφορετικά στοιχεία τα οποία ε, έπρεπε να ληφθούν υπόψη όταν ξεκινήσαμε την κίνηση προς μια τραπεζική ένωση. Ξέρω τώρα βέβαια ότι υπάρχει το θέμα του κρατικού χρέους. Αναρωτιέμαι αν αυτό είναι η μόνη πηγή κινδύνου, θα ήθελα να ξέρω και την άποψή σα για το πώς θα πρέπει να ε, υπολογίζετε την κεφαλαιοχική επάρκεια, αν υπάρχει επαρκή διαφάνεια για τα θέματα αυτά. Και τον κύριο Τανιέλ Κρός, σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ. Και το ερώτημά μου έχει να κάνει περισσότερο με το γεγονός ότι φαίνεται να συμβάλλετε με ένα νέο στοιχείο στην θεματολογία όταν λέτε ότι οι μικρές τράπεζες και οι μεγάλες τράπεζες πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Εσείς θεωρείτε ότι κατά πόσα πιθανότητα οι μικρές τράπεζες δεν θα πρέπει να συμβάλλουν σε ένα κοινό ταμείο επίλυσης και να έχουν απλώς εθνικά συστήματα επίλυσης που να περιλαμβάνουν και το σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Γιατί αν είναι στο ίδιο σύστημα ε, εποπτείας και συμβάλλουν στο ίδιο σύστημα εγγύησης καταθέτων, θα πρέπει να καλύπτονται με τον ίδιο τρόπο οι καταθέσεις σε όλες τις ε, τράπεζες σε όλες τις χώρες που υπόκεινται στην Τραπεζική Ένωση. Στην κυρία Κιόνιχ, νομίζω ότι είναι σημαντικό όταν συγκρίνεται την κατάσταση στην Ευρώπη με το Αμερικανικό σύστημα, το FDIC. Στην αρχή αυτό ήταν στο μυαλό μας να βρούμε ένα σύστημα το οποίο θα μπορεί να αντιμετωπίσει μια συστημική κρίση όπως οι ΗΠΑ. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι να έχουμε αυτή την αρχική ιδέα ενός συστήματος που θα, ήταν, είχε, θα είχε ομοιότητες με το FDIC. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και όλους τους ομιλητές. Εάν κατάλαβα καλά, ο κύριος Γκρός είπε στο τέλος της ε, παρέμβασής του ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ένα σύστημα ε, εγγύησης παρεμβαίνοντα σε ελάχιστο επίπεδο στι εθνικέ ε, αρμοδιότητε. Είπατε προηγουμένω, κύριε Βούλφ, να αναφέρεστε στο γεγονό ότι τα κράτη-μέλη ακόμα αποφασίζουν για τι εθνικέ οικονομικέ και δημοσιονομικέ πολιτικέ, οι οποίε φυσικά επηρεάσουν και τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών. Μήπω θα μπορούσατε να πείτε κάτι περισσότερο, με ποιο τρόπο μπορούμε να έχουμε ένα πλήρε σύστημα ε, ευρωπαϊκής ε, γη καταθέσεων που να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, καθώς και τον ηθικό κίνδυνο που προκύπτει από το γεγονός ότι παραμένουν εθνικές αρμοδιότητες. Έχουμε μεγάλες επίσης διαφορές στο εθνικό πτωχευτικό δίκτυο και επίσης να ρωτήσουμε στην κυρία Κιόνιχ είπατε προηγουμένως και δώσατε αυτό το κέριο μήνυμά σα, το οποίο ανέφερε και η κυρία Φερέιρα, ότι πρέπει να υπάρξει και μια λύση για τις μικρές τράπεζες. Έχουμε πει πάρα πολλά για τις ε, συμβολές που θα πρέπει να δοθούν από τι τράπεζες στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων, το αναφέρει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην γνωμοδότηση που είχε δώσει για την πρόταση για το σύστημα EDIS. Το ερώτημα είναι πρέπει οι μικρές τράπεζες να πληρώνουν αναλογικά περισσότερο γιατί είναι πιο πιθανό να δημιουργηθεί κάποια ανάγκη αποσημείωσης καταθετών. Ποια είναι η απόψη σε αυτό το σημείο. Ευχαριστώ. Η Σιλβί Γκουλάρ. Ευχαριστώ πολύ σας, ευχαριστώ όλους για τη συμβολή σας. Έχουν τεθεί πολλά ερωτήματα, εγώ θέλω απλώς να σταθώ σε δύο σημεία που μου φαίνονται σημαντικά. Πρώτον, θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψή σας σε σχέση με τον αντίκτυπο μεταξύ των τραπεζών της ζώνης του ευρώ και των τραπεζών που είναι εκτός της ζώνης του ευρώ, γιατί σε επίπεδο Ευρωπαϊκή, Ευρώπης 28 θα πρέπει να έχουμε ισότητα ανταγωνισμού. Και ήθελα να ρωτήσω τον Κούντραν Βόλφ τι εννοεί όταν λέει μια ισχυρή νομική βάση λέτε ότι δεν πρέπει να παραμείνουμε μέσα στις συνθήκες και να ξαναμπούμε στην ε, περιπέτεια στην οποία μπήκαμε με την ε, τραπεζική επίλυση ή πρέπει να παραμείνουμε στα πλαίσια των συνθήκων. Ποια είναι η ισχυρή νομική βάση με την οποία καταφέραμε να κρατήσουμε ή να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Παπαδημούλης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους ομιλητές για τη συμβολή τους να τους δώσω και λίγα δευτερόλεπτα για να χρησιμοποιήσουν ακουστικά όσοι δεν έχουν και να ρωτήσω τα εξής. Ε, καταρχήν να πω ότι με εντυπωσίασε η ισχυρή σύγκληση των απόψεων των ειδικών. Διαπιστώνω ότι είναι ισχυρότερη από τη σύγκληση που μέχρι στιγμής έχουμε εμείς στο Κοινοβούλιο σε ένα θετικό πνεύμα ότι χρειάζεται να προχωρήσει και ο τρίτος πυλώνας. Η ερώτησή μου είναι και προς τους τέσσερις πότε νομίζετε ότι πρέπει να αρχίσει να δουλεύει αυτό που περιγράψατε. Έχουμε πολλά χρόνια μπροστά μας που μπορούμε να καθυστερούμε και να αναβάλουμε. Και επίσης ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κουπέ η γνώμη σας για την πρόταση που έχει καταθέσει η Κομισιόν καταρχήν είναι θετική ή αρνητική δεν κατάλαβα. Για τους άλλους τρεις ομιλητές είδα ότι το προσεγγίζουν το θέμα θετικά. Η δική σας γνώμη ποια είναι. Είστε καταρχήν υπέρ και μια, μια ερώτηση και προς τους τέσσερις. Αν σας ζητούσαν ε, να προτείνετε ένα-δυο πράγματα, τα πιο βασικά κατά τη γνώμη σας, που πρέπει να προσεχθούν ή να αλλάξουν στην πρόταση που έχει καταθέσει η Κομισιόν. Ποια θα ήταν αυτά. Ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ, Φίλιπ Λεμπέτς. Καλησπέρα σε όλους. Η δικιά μου ερώτηση απευθύνεται στον, στους Γκούντραμ και Ντανιέλ. Ένας τρόπος ε, για να μειωθεί αυτό το πλέγμα κρατών ε, και τραπεζών ε, και ο κίνδυνος ταυτόχρονα είναι να υπάρξει μία μεγαλύτερη ποικιλομορφία όσον αφορά το χρέο στα κρατικά ομόλογα. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε στι τελικέ τράπεζε δεν θα έχετε πολύ μεγάλο τελικό χρέο ή αλλιώ να ενθαρρύνουμε κάθε δανειστή στην Ευρώπη ε, να έχει ένα χαρτοφυλάκιο δημοσίου χρέους από πολλές ε, πηγές, ε, κάτι το οποίο βεβαίως σημαίνει ότι θα αυξανόταν το... αλλά και θα μοιραζόταν το ρίσκο για τους δανειστές και για τα κράτη. Ποια θα ήταν η απόψή σας για κάτι τέτοιο, με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και για την κυρία Κένιγκ. Αντιλαμβάνομαι ότι στον πρώτο μιλτή δεν αρέσει το σύστημα, οπότε Ναι, φαντάζομαι πως κάτι τέτοιο θα απαιτούσε κάποιο στοιχείο το οποίο θα ήταν τελείως ελεύθερο από κείμενο. Λοιπόν, Χάνεμανς. Ε, ε, Ευχαριστώ. Νομίζω πως ε, μπορεί ο κάθε ομιλητής να κρίνει αν θέλει να απαντήσει ή όχι. Ε, εδώ πέρα βλέπω μια παλιά αναφορά του κυρίου Γκρός για έναν όγκο 55 δισεκατομμύρια. Γιατί ποσά ακριβώς ε, μιλάμε. Αν σκεφτούμε ότι το Βέλγιο είχε χρειαστεί γύρω στα 20 δισεκατομμύρια, δεν νομίζω να υπάρχει. Έχετε κάποια ιδέα λοιπόν για το ποσά τα οποία μιλάμε. Και δεύτερον, ένας, κριτικής έκανε ένας ομιλητής έκανε κάποια κριτική, δεν ξέρω αν θα ήθελαν και οι άλλοι να επανέλθουν, για το νομικό πλαίσιο. Εμείς θα το παρακολουθήσουμε και οπωσδήποτε θα παρεμβούμε στην ε, διαδικασία αυτή γιατί θεωρούμε ότι ξεπερνά τα όρια και κινούμαστε σε μια γκρίζα ζώνη τι άποψη έχετε, είναι ρεαλιστικό κάτι τέτοιο ή όχι. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε και τώρα διαδικασία. Κάτσε, δια, κύριος Τσέκερ πρώτος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία συγκεκριμένη ερώτηση προς τον Ντανιέλ. Ναι, καταλαβαίνω ότι πόσο είναι θετική η αντασφάλιση που προσφέρει κάποια πλεονεκτήματα. Όμω, επισημαίνω δύο προβλήματα και περιμένω πώ και πώ να μου απαντήσει πρωτα πρώτα-πρώτα. Δεν έχουμε κάποιο είδου ε, ε, χρηματοδοτικό backstop και δεν έχουμε και στο σύστημα αντασφάλισης. Επομένως, δεν ξέρω, θα έχουμε τέτοιου η είδους σύστημα αντασφάλισης όπως ε, ε, ανέφεστο ώστε να δημιουργήσουμε με αυτό το backstop, με αυτή τη στήριξη ασφάλεια, την δημιουργία εμπιστοσύνης. Επίσης θα πρέπει ό,τι σχεδιάζεται να είναι επί τη βάση της εκτίμηση του κινδύνου. Έχεις ε, στα θέματα κοινότητας εμπειρία. Οπότε πόσο ρεαλιστικό θα είναι να έχουμε ένα τέτοιο σύστημα ε, εισφορών αυτής τη αντασφάλισης που να βασίζεται στην εκτίμηση του κινδύνου γιατί είναι βάσιμο το επιχείρημα αυτό για το σύστημα ασφάλισης. Ευχαριστώ, Πίτερ Τζίμαν. Εγώ θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα για την τελική φάση, την τελευταία φάση και την κατάσταση που θα δημιουργηθεί όταν έχει ουσιαστικά αδειάσει το ταμείο από τις σύμβολες των τραπεζών. Πώς θα υπάρξει η επανα ε, αυτού του ταμείου με τη βάση ποιων παραμέτρων θα γίνει αυτό ε, όταν υπάρχει ανάγκη να καλυφθούν πάλι τα ποσά αυτού του ταμείου το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί για κάποια συγκεκριμένη αντιμετώπιση ενός προβλήματος. Και αν λάβετε υπόψη το γεγονός ότι μια τράπεζα μπορεί να βρίσκεται σε δυσκολία λόγω συστημικών ε, παραγόντων, δεν υπάρχει ο κίνδυνος μια ομάδα τραπεζών να βρίσκεται συνέχεια στην ανάγκη να δίνει συμβολές σε αυτό το ταμείο. Πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό το κίνδυνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Δεν βλέπω στα πλαίσια του κάτι άλλο ζητεί το λόγο. Επομένως τώρα να στραφώ στους προσκεκλημένους μας για να απαντήσουν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λέω κύριε Σκουπάη, το, ε, επί τη βάση όσων ρωτήσατε για το πώς ε, αυτό το σύστημα θα καλύψει τα διάφορα προβλήματα, για τα διάφορα συστήματα εγκυοδοσίας. Σε σχέση με σου κυρία Κιονίκη, θα πρέπει η οδηγία να μεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο όλων των κρατών μελών. Σου και νέος κανονισμός. Αυτό το επικρίνουμε πάντα ότι θα πρέπει όλη αυτή η νομοθεσία να εφαρμοστεί στα κράτη-μέλη. Να υπάρχει δηλαδή μια τέτοια δομή εγγυητική. Πάντως πλησιάζουμε και επικυροποιούμε την ενημέρωση των κρατών μελών για όλα τα συστήματα που υπάρχουν. Άρα να μην υπάρχει φάση μεταφοράς, να εφαρμοστεί απευθείας και αυτή η ασφάλιση των καταθέσεων να μην έχει ε, μεγάλες φάσεις αποπληρωμής. Αυτό το οποίο θέλουμε να δούμε τι εναλλακτικά μέτρα μπορεί να έχουμε πριν την παρέμβαση του Ταμείου αυτής της ε, ασφάλισης και υπάρχουν διαφορές μεταξύ των εθνικών συστημάτων. Φτάνουν μέχρι το 0,8% όσον αφορά την ε, κάλυψη των τραπεζών. Θα πρέπει να δούμε πώς θα ελαφρώσουμε το βάρος στο εθνικό τραπεζικό σύστημα. Να δούμε τι βοήθεια έχει δοθεί σε κάποια τράπεζα εκ των προτέρων πριν έρθει η ώρα ε, της εφαρμογής του συστήματος εξασφάλισης. για κάποια pay boxes έχουμε άλλη ρύθμιση και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε στην ε, υλοποίηση και εφαρμογή αυτής της ε, οδηγίας και πώς έχουν τα πράγματα σε αυτήν την περίπτωση. Η κυρία Γκουλάρ μας μίλησε για την νομική βάση. Εμείς λέμε ότι έχουμε το άρθρο 352 αυτό θα μπορούσε να είναι η νομική βάση. Όπως έγινε και με τις διακυβερνήσεις μας για το SRB και SM, πάντως υπάρχουν και κάποιες ε, σοβαρές αμφισβητήσεις. Επίσης, πόσο θα μας πάρει να καταφέρουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Θα εξαρτηθεί πόσο θα, θα συζητήσουν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για να καταλήγουν σε ένα τελικό μοντέλο. θα χρειαστεί κάποιο χρόνο, πιστεύω. Γιατί νομίζω ότι οι ασφαλείς μεταθέσεων είναι βασικό εργαλείο για το τραπεζικό σύστημα. Έχουμε φτάσει στην τελική φάση, αλλά τώρα έχουμε διάφορε προποθέσει που θα πρέπει να συντρέξουν. Να δούμε και το πώ θα μειώσουμε του κινδύνου, μελέτη των επιπτώσεων. Θα πρέπει να δούμε κάποια πράγματα ε, παραπάνω. Γιατί είπαμε η τάση είναι να έχουμε τελικά ένα σύστημα που να καλύπτει όλη την Ένωση και όχι μόνο την Ευρωζώνη. Ο κύριος ε, Χάνομανς μας είπατε για αυτά τα 20 ε, δις, ε, αλλά δεν μιλάμε το. Μιλάμε τώρα για διάσωση, για εξυγίανση. Ας πούμε τι έγινε με την φόρτη στο Βέλγιο. Τώρα έχουμε διαφορετικό σύστημα ε, διάσωση και μιλούσαμε για ρευστότητα και όχι για ζημία σε εκείνη την περίπτωση. Τώρα θα πρέπει να δούμε το ότι πέρσι, τον Σεπτέμβριο, είχαμε κάποια στοιχεία για τις καταθέσεις. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015 κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει όμως αυτός ο στόχος του 0,8% αν ισχύει για μια χώρα τη Ευρωζώνης ή για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν υπήρχαν στοιχεία για κάλυψη καταθέσεων και μόλι τον Σεπτέμβριο. Για πρώτη φορά είδαμε κάποια στοιχεία, οπότε είδαμε πώς μπορεί να υπολογιστεί το τι θα γίνει για να φτάσουμε ε, στην καταλητική μερία του 2024 που είναι σαν προθεσμία αυτής της ε, νομοθετικής πρότασης με κύριο Τζίμαν ναι, είπαμε ότι θα πρέπει η χρηματοδότηση να γίνεται εκ των προτέρων. Δεν μπορεί κανεί να δεσμευθεί από τον προτέρων για το πόσα θα χρηματοδοτήσει. Θα πρέπει επομένω να καλυφθούν και οι ζημίε. Αλλά θα πρέπει επίση να υπάρξει μια ε, χρηματοδότηση για τις καθημερινές ε, ανάγκες και θα πρέπει ό,τι προβλεφθεί να είναι ξεκάθαρο και διάφανο για όλους. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ για την απάντηση κύριε Κούπε. Αλλά δεν νομίζω ότι σας τα ερώτησα τόσο ξεκάθαρα. Αν μπορείτε, πέστε μας τι ισχύει σήμερα. Γιατί όσον αφορά την μεταφορά στο ιστορικό δικαίο, εγώ έχω απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα, όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, πώς λειτουργούν τα επιμέρους εθνικά συστήματα, ποιος είναι ο βαθμός διαφάνειας Και στα πλαίσια της Τραπεζικής Ένωσης η σύγκριση τι μας δείχνει. Με μεγάλη χαρά μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένα στοιχεία για τα θέματα αυτά και πάντα εμείς τα επικαιροποιούμε αυτά όταν έχουμε νέα με, με λύκη ή όταν αλλάζουν οι εθνικές νομικές βάσεις. Έχουμε λοιπόν συστήματα που είναι ιδιωτικά, είναι εθνικά, είναι μεικτά, έχουμε συστήματα από τη βάση συμβολών, έχουμε συστήματα που έχουν συγκεκριμένους στόχους. Είναι τόσο ετερογενή λοιπόν και διαφορετικά τα συστήματα τώρα που είναι πολύ δύσκολο εδώ σε λίγα λεφτά να σας εξηγήσω ποιε είναι οι διαφορές των εθνικών συστημάτων. Είναι πολύ λοιπόν ε, διαφορετικά τα συστήματα αυτά. Υπάρχει τώρα η οδηγία αυτή για την εγγύηση των καταθέσεων η οποία θα εφαρμοστεί βέβαια. Θα σας δώσω λεπτομέρειες για όλα τα συστήματα των 28 χωρών και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ένωσης. Επίσης, ευχαριστώ, Αντέο ο Κάτι το οποίο είναι σαφές και σίγουρο είναι ότι για, ένα κοινο, για το κοινοβουλίο μας μια διακυβερνητική συμφωνία δεν θεωρείται ότι είναι ισχυρή νομική βάση. Ο κύριος Βόλφ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Εννέα ερωτήσεις μου απευθύνανε και νομίζω ότι έχω έχω τρία-τέσσερα λεπτά. Θα προσπαθήσω να τις ομαδοποιήσω λιγάκι. Το πρώτο θέμα είναι τι γίνεται με τις τράπεζες που είναι στην Ευρωζώνη και αυτές που είναι εκτός. Υπάρχει μια διαφορετική λογική. Υπάρχει μια λογική νομισματικής και οικονομικής ένωσης και υπάρχει και η νομική η, η, συγνώμη, η νοοτροπία της ε, Τραπεζικής Ένωσης. Όλα ξεκίνησαν από την Νομισματική Ένωση βέβαια γιατί είχαμε μια μεγάλη κρίση αλλά όταν θέλουμε να έχουμε μια, μια ε, τραπεζική ένωση για τις χώρες του ευρώ, δημιουργείται μια μεγάλη στρέβλωση για τις χώρες που είναι εκτός. Αν μονάχα υπάρχει λοιπόν εγγύηση καταθέσεων για την περιοχή του ευρώ, αυτό θα έχει επιπτώσεις για τις, περιοχές που, για τις χώρες που δεν είναι μέσα στη ζώνη του ευρώ. Αυτό συμβαίνει ήδη και με την νομισματική ένωση. Από τη στιγμή που υπάρχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η πρόσβαση στη ρευστότητα, η αξιοπιστία των τραπεζών επηρεάζεται ήδη ακόμα και για τις χώρες εκτός της νομισματικής ένωσης. Το δεύτερο ερώτημα τώρα αφορά σε ποιο βαθμό πρέπει να προχωρήσει η εναρμόνιση, μέχρι πού μπορούμε να πάμε, αν μπορούμε να διατηρήσουμε την ε, εθνική ε, διακριτική ευχέρεια, παραδείγματος χάρη στο πτωχευτικό δίκαιο κτλ. Εγώ νομίζω ότι για μένα είναι σαφή τα πράγματα. Αν θέλετε απόλυτα να αποσυνδεθούν οι τράπεζες από, ε, από το κρατικό χρέο, θα πρέπει να υπάρξει το πλήρε σύστημα ευρωπαϊκή ασφάλεια καταθέσεων. Αλλά δεν μπορείτε να το έχετε αυτό χωρί να υπάρξει και εναρμόνιση στη λειτουργία της εγγύησης καταθέσεων. Αυτό πάει μακριά. Αν η πολιτική εκτίμηση είναι ότι πρέπει να διατηρηθούν κάποιες διακριτικές ευκαιρίες σε εθνικό επίπεδο, παραδείγματος χάρη η διαφορετική αντιμετώπιση των ε, ε, καταθέσεων όταν κανείς θέλει να αγοράσει ένα σπίτι και εκεί πέρα πρέπει να ξεπερνάει κανείς το όριο των 100.000 ευρώ. Αν έχετε λοιπόν μονάχα ένα σύστημα, ένα ευρωπαϊκό ενίο σύστημα, δημιουργούνται δυσκολίες γιατί δεν καλύπτονται όλες αυτές τις περιπτώσεις. Γι' αυτό εγώ εξέφρασα μεγάλη κατανόηση για το μοντέλο αντασφάλισης που ανέφερε ο Ντάνιελ Γκρός. Διατηρεί ε, το στοιχείο της ε, επικουρικότητας και επιτρέπει σε ένα ε, επίπεδο που είναι κάτω από το ανώτερο επίπεδο να διατηρούνται οι ιδιαίτερες των κατωμένων, αλλά με τον τρόπο αυτό δεν θα αποσυνδέσετε τις τράπεζες από το κρατικό χρέος και θα διατηρήσετε κάποια σύνδεση σε ορισμένε χώρες. Αν είναι το κρατικό χρέο ο μόνος κίνδυνο, όχι βέβαια, υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι. Το ερώτημα είναι πόσο εξαρτώνται οι άλλοι κίνδυνοι από τις εθνικές πολιτικέ, Βεβαίως εξαρτώνται, αλλά το πραγματικό ερώτημα είναι αν υπάρχει μια θεληματική πολιτική ώστε κάποιος να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εγγύησεων ακόμα και στην πιο ακραία κατάσταση που είχαμε πέρσι στην κρίση στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι κανείς ήθελε στην Ελλάδα να υπάρξει ε, μαζική απόσυρση ε, από τους καταθέτες στις ελληνικές τράπεζες. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν του ηθικού κινδύνου ότι το σύστημα εγγυήσεων μπορεί να οδηγήσει σε μαζική απόσυρση από τους καταθέτες, αυτό πραγματικά δεν νομίζω ότι ευσταθεί θα πρέπει να είμαστε κάπως πιο καθυσχασμένοι για το θέμα αυτό. Ένα από τα βασικά προβλήματα είναι ακριβώς όμως αυτά τα κρατικά ομόλογα που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο των τραπεζών και εδώ πιστεύω ότι υπάρχει πάλι μια ασυνέπεια αν θέλετε αν υπάρχει σημαντικό εθνικό χρέος στο χαρτοφυλάκιο μιας τράπεζας και έχετε μια τράπεζα η οποία χρηματοδοτείται κυρίως από τους καταθέτες και έχει ένα μικρό μετοχικό κεφάλαιο και έχει στα βιβλία της κυρίως εθνικό χρέος. Τότε ουσιαστικά με το σύστημα ασφαλίσεως ε, καλύπτεται τις απώλειες που μπορούν να προκύψουν από ε, μείωση της αξίας του εθνικού χρέους και αυτό θα πρέπει να καλυφθεί από το σύστημα εγγύησεως. Αυτό είναι ένα πρόβλημα όσο οι δημοσιονομικές πολιτικές είναι ακόμα εθνικού χαρακτήρα. Γι' αυτό έχουμε το εργαλείο τελικής καταφυγής να γίνεται το bail-in για το κρατικό χρέος. Η συμμετοχή λοιπόν των καθατεθωτών και ομολογιούχων. Αυτό είναι ένα ακραίο μέτρο το οποίο είναι δυσάρεστο, δεν γίνεται πολύ συχνά και ιδανικά δεν θα πρέπει να γίνεται ποτέ. Όσο όμως έχουμε ακόμα κεντρική νομισματική πολιτική και αποκεντρωμένη δημοσιονομική πολιτική πάντα θα έχετε τέτοια προβλήματα. Και έρχομαι τώρα στο ερώτημα του κύριου Λάμπερτ για την ε, διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων των τραπεζών. Όσο έχουμε λοιπόν αυτό το σύστημα, σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη διαφοροποίηση και το κρατικό χρέος να κατανέμεται σε όλη την Ευρωζώνη. Μια ενδιαφέρουσα επιλογή θα ήταν να πείτε ότι δεν υπάρχει θεωρείται ότι είναι μηδενικού κινδύνου το χαρτοφυλάκιο μια τράπεζα αν έχει μια ποικιλία κρατικών ομολόγων, όχι μόνο από τη δική τη χώρα, αλλά και από άλλε χώρε. Υπάρχει βέβαια ο κίνδυνο για το κρατικό χρέο, αλλά υπάρχει μια διαφορετική σύνθεση του χαρτοφυλακίου για την νομική βάση. Δεν είμαι πυρογνώμο στα νομικά, Σιλβί. Αλλά άμα κάνετε κάτι το οποίο δεν έχει μια ισχυρή νομική βάση και υπάρξει μια κρίση, τότε φτάνετε στα δικαστήρια και εκεί πέρα όχι μόνο έχετε ένα πρόβλημα, αλλά χάνετε και κάθε αξιοπιστία. Προφανώς χρειάζεστε μια ισχυρή νομική βάση και πολλοί λένε ότι το άρθρο 114 δεν επαρκεί, ιδίω άμα καλύπτει μονάχα ρυθμίσει στην Ευρωζώνη. Και αυτό είναι θέμα, αλλά και πάλι πηγαίνετε στου δικηγόρου τώρα πώ πρέπει να αναπληρώνετε το ταμείο όταν εξαντληθεί. Αν υπάρξει ένα μεγάλο πληρονισμό θα πρέπει να ε, αναπληρωθεί με τέλη τα οποία επιβάλλονται στις καταθέσεις. Αλλά αυτό είναι κάτι που πρέπει να αποφασίσουν οι δύο στις τράπεζες. Ευχαριστώ. Ντάνιελ έχει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ομοδοποιήσω λίγο τις ε, ερωτήσεις. Ποια είναι η κυριότερη αλλαγή την οποία θα ήθελα. Απλό η φάση της αντασφάλισης να μην είναι φάση αλλά να είναι μόνιμη. Για το θέμα τώρα της, ε, του αμοιβαίου δανεισμού και αν επαρκεί σε ένα μεγάλο σοκ, η απάντησή μου θα είναι πως ε, όταν καίγεται το σπίτι σου δεν χρειάζεσαι δάνειο από το γείτονα, αλλά από την ασφαλιστική εταιρεία για να το ξαναφτιάξεις. Οπότε στην περίπτωση ενός ε, μεγάλου σοκ οι υπόλοιποι θα πούν θέμα να δανείσουμε, οπότε αμοιβαίος δανεισμός δεν αρκεί. Για τις μικρές τράπεζες είναι αυτές στις οποίες ο παρακαθήμενος εδώ πέρα βεβαίως δεν θα ασχοληθεί τόσο πολύ, αλλά θα πρέπει βεβαίως και οι δικοί τους καταθέτες να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Αλλά νομίζω πως μπορούν να να αντιμετωπιστούν από τα εθνικά συστήματα και είναι αυτά τα οποία παρέχουν εποπτεία ούτως ή άλλως και μπορούν να κρίνουν καλύτερα από κάποιον ο οποίος βρίσκεται στην Φραγκφούρτη, ειδικά για τις μικρές τράπεζες, ε, ποιο είναι ο κίνδυνος της ε, κάθε τράπεζας. Οπότε μπορούν να μείνουν στο εθνικό επίπεδο και οι μικρές τράπεζες ε, δεν ε, οδηγούν και σε αυτόν τον φαύλο κύκλο μετά μεταξύ τραπεζών και κρατών. Μετά, το θέμα του εάν η αντασφάλιση αυτή θέτει ιδιαίτερα προβλήματα και για το θέμα του δημοσιονομικού αυτού αποθεματικού και των ε, εισφορών. Είτε ακολουθήσουμε λοιπόν ε, την ανασφάλιση είτε όχι, ε, τίστε το ζήτημα. Δεν υπάρχει λοιπόν ιδιαίτερο πρόβλημα με την προσέγγιση της ανασφάλισης για τις εισφορές με βάση τον κίνδυνο. Νομίζω πως η πραγματικότητα έχει δείξει στην περίπτωση του FRF πως αν πάμε σε μια διακυβερνητική προσέγγιση, η ψαλίδα μεταξύ των εισφορών είναι κάπως μικρή, καθώς ε, κάθε χώρα προσέρχεται στις διαπραγματεύσεις με ένα στόχο, να γλιτώσει λεφτά. Αλλά βεβαίως, ε, εντάξει, στο σύνολο μετά δεν μπορούν όλοι να γλιτώσουν λεφτά, οπότε συνήθως ε, ο ελάχιστος κοινό παρανομαστής μετά είναι πάρα πολύ μικρές εισφορές με βάση τον κίνδυνο. Εγώ θα έλεγα πως στην προσέγγιση της αντασφάλισης. Μπορεί να υπάρχει κάποιος αντασφαλιστής ο οποίος θα έχει περισσότερο ένα σχήμα ομοσπονδιακό και λιγότερο διακυβερνητικό και άρα θα υπάρχει ακριβώς και αυτή η διαφοροποίηση με βάση το ρίσκο που είναι θα έλεγα περισσότερο μακροοικονομικός ο κίνδυνος αυτός. Το ζήτημα είναι το ποιες θα είναι οι εισφορέ που θα πληρώνει το εθνικό σύστημα στο ομοσπονδιακό μαζί σε συνδυασμό με τη μακροοικονομική κατάσταση με τη διαδικασία δηλαδή υπερβολικών ανισορροπιών που μα δίνει μια ιδέα του πόσο μεγάλος ε, είναι ο κίνδυνος ενό συστημικού σοκ στο εθνικό επίπεδο και αντί να παρεμβαίνει η Κομισιόν με πρόστιμα θα μπορούσε να συνδεθεί με ακριβώς ε, την ευρωπαϊκή αντασφάλιση που είναι μια εναλλακτική στα πρόστιμα ή στις ε, αποφάσεις του Συμβουλίου. Είναι μια κάπως πιο διαφοροποιημένη αντίδραση. Οπότε η προσέγγιση της αντασφάλισης για μένα έχει και άλλα δύο επιπρόσθετα πλεονεκτήματα. Θα έλεγα πως μπορεί να εφαρμοστεί πιο γρήγορα, γιατί μπορεί να βασίζεται στο υφιστάμενο εθνικό επίπεδο και θα επιτρέπει την διαφοροποίηση που ανέφερε ο Γκούρτραμ, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε ευθύ αμέσω χωρίς ε, να υπάρχει εναρμόνιση των πάντων, ειδικά όσον αφορά την εναρμόνιση του πτωχευτικού δικαίου. Μπορούμε να εναρμονίσουμε το δίκαιο, αλλά το αποτέλεσμα, οι διαδικασίες ε, δεν εναρμονίζονται αρκεί να δούμε στην Ιταλία όπου είναι ίδια η νομοθεσία, πόσο χρειάζεται ίδια διαδικασία στο Μιλάνο και στο Παλέρμο. Τα ξέρει και ο κύριος Πρόεδρος. Είναι το θέμα της εφαρμογής λοιπόν, όχι μόνο του δικαίου. Και τέλος, ε, η διαφορά μεταξύ μιας προσέγγισης ε, με τα που θα είναι μόνο στην Ευρωζώνη ή σε όλα τα κράτη-μέλη αποκτά λιγότερη σημασία γιατί ακόμα και χώρα που δεν είναι στην Τραπεζική Ένωση θα βλέπει ότι υπάρχει συμφέρον στην αντασφάλιση στην περίπτωση που υποστεί πίεση το δικό της ε, τραπεζικό σύστημα. Και ακριβώς υπάρχει αυτή η διαφορά μεταξύ Ευρωζώνης και Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία με την αντασφάλιση θα αμβλυνθεί. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Κένιγκ, σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λάγκη δεν μπόρεσε να αντισταθεί για το τίλεκ και εγώ δεν μπορώ να αντισταθώ στο να απαντήσω. Για μένα το Emerald είναι βασικό γιατί είναι το εργαλείο που έχει το Συμβουλίο Συνδική Σταθερότητα και ο Μηχανισμός Διάσωσης για να διασφαλίσουμε ότι οι τράπεζες, οι μεγάλες τράπεζες λέμε εδώ πέρα που μα αφορούν εμά, έχουν τη δυνατότητα να διασωθούν και υπάρχουν τα σχετικά κίνητρα. Και εμείς πάντα λέμε πως δεν βλέπουμε ανάγκη να αλλάξει η άποψή μας. Ότι δηλαδή το 8% ή και για κάποιες τράπεζες ακόμη περισσότερο, για τις μεγάλες τράπεζες στην Τραπεζική Ένωση, είναι μια καλή αφετηρία για να βασιστούμε ποσοτικά. Η ποιότητα μετά είναι κάτι το διαφορετικό. Θα σταματήσω. Λοιπόν, οι ερωτήσεις αφορούσαν το τι θεωρούμε ότι θα... ποια είναι η κύρια αλλαγή που χρειάζεται. Άκουσα πολύ προσεκτικά τα όσα είπε ο Γκρός για την αντασφάλιση και οι εισφορές με βάση τον κείμενο είναι οπωσδήποτε μια πολύ καλή αρχή. Αλλά για μένα το βασικό είναι να έχουμε ένα σύστημα που θα κάνει την δουλειά του, που θα περιλαμβάνει και τα εναλλακτικά μέτρα. Και αυτή ήταν νομίζω η ερώτηση της κυρίας Φερέρα, δηλαδή ποια είναι τα μαθήματα που αντλούμε Κοιτάξτε, να σκεφτούμε ότι το αμερικανικό σύστημα έχει εμπειρία 80 ετών. Οπωσδήποτε η εμπειρία τους ε, είναι ότι μεταφέρουν τους ε, καταθέτες σε ένα άλλο ίδρυμα. Και αυτός είναι ο πιο αποτελεσματικός ε, τρόπος να μην έχουν πρόσβαση μετά από 7 μέρες, αλλά να υπάρχει ε, άμεση πρόσβαση στις ε, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες για τους πελάτες. Για μένα αυτό είναι νομίζω ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, είτε ε, ευρωπαϊκό είτε εθνικό σε ένα σύστημα αντασφάλισης. Και βεβαίως το θέμα της εναρμόνισης του πτωχευτικού δικαίου και των διαδικασιών πολύ περισσότερο. Για να επανέλθω λοιπόν στις άλλες ε, ερωτήσεις. Η λύση για τις μικρότερες τράπεζες σε σχέση με τις μεγαλύτερες. Ε, όπως το βλέπω εγώ. Στις ε, περισσότερες περιπτώσεις που ελπίζουμε να μην συμβεί για ένα μεγάλο ίδρυμα με στιβαρό έμπρελ, δηλαδή με χρέος ε, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσουμε για μπέιλιν και με ένα ενιαίο ταμείο διάσωσης δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να εκτεθεί το σύστημα ασφάλισης καταθέσεων σε μεγάλες απώλειες. Στην περίπτωση αυτή δεν θα μιλάμε μάλλον για κρίσιμες λειτουργίες και για την ε, χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ενίας αγοράς ή ενός ολόκληρου κράτους μέλους. Εδώ πέρα λοιπόν η πρώτη γραμμή άμυνας είναι το σύστημα εγγύηση καταθέσεων για να μην υπάρχουν και άνηση όροι ανταγωνισμού καθώ οι μεγαλύτερες τράπεζες ε, θα θεωρούνται τότε πιο ασφαλείς. Και το συνδέσατε και με το ποιο θα πρέπει να πληρώνει περισσότερο. Εγώ θα έλεγα πως και οι δύο πρέπει να πληρώνουν το ίδιο. Αυτοί οι οποίοι πιθανώς δεν θα έχουν πρόσβαση ποτέ, θα πρέπει να πληρώσουν γιατί έτσι υπάρχει περισσότερη σταθερότητα στο σύστημα και τότε γιατί να μην κάνουμε το αντίστροφο και να πληρώσουν όλες οι τράπεζες γιατί έτσι υπάρχει ε, περισσότερη εμπιστοσύνη και σταθερότητα στο σύστημα. Τώρα για την διαφοροποίηση του δημοσίου χρέους εγώ πάντα θεωρούσα πως ε, το ότι δεν υπάρχει κάτι χωρίς κίνδυνο, αλλά η απάντηση βεβαίως είναι πολύ πιο περίπλοκη εδώ πέρα και αφορά την μείωση του κινδύνου. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να υπάρξουν κάποια όρια συγκέντρωσης, ε, αλλά να μην λέμε ποιος θα επενδύσει τι. Το άλλο ερώτημα ήταν ποιο ήταν το ύψος, γιατί ποσά μιλάμε και πώς θα γεμίσει, θα έλεγα, το ταμείο αυτό. Πράγματι πρέπει να υπάρχει μια αντίληψη του πώς θα ξαναγεμίσει αυτή τη στιγμή σε χρησιμοποιηθεί. Λοιπόν, για το ύψος 1% των καλυπτόμενων καταθέσεων είναι το σημείο αναφοράς ε, για το Ταμείο Διάσωσης. Ένα 0,8% θα έλεγα πως είναι μια καλή αφετηρία για την εγγύηση των καταθέσεων και μετά βλέπουμε. Και θα πρέπει βεβαίως ε, να δούμε το τι γίνεται και αλλού ε, στο ενιαίο Ταμείο Διάσωσης για το πώς θα ξαναγεμίσει το Ταμείο αυτή τη στιγμή χρησιμοποιηθεί γιατί μπορεί να συμπέσουν κάποια γεγονότα και να υπάρχει όριο στην αναχρηματοδότηση. Ε, σίγουρα κάποια πράγματα παρέλειψα, αλλά θα σταματήσω εδώ. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ήταν αυτό το πρώτο μέρος ακρόασης και τώρα πάμε στο δεύτερο να δούμε το τι διεύματα πρέπει να γίνουν μέχρι την τελική φάση. Ε, βεβαίως ε, τα προηγούμενα και τα επόμενα αλληλοσυνδέονται. Τώρα η κυρία Ρόζμπεκ από την ΣΥΠ, ε, e από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Έλληνα, έχετε το λόγο. Ο κύριο Φανερόζμπεκ, ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστούμε. Καλέσατε, μου δώσατε δυνατότητα να σα τα πω σήμερα σε σχέση με ε, αυτό το σύστημα ασφαλή καταθέσεων. Μπορώ να προσθέσω μερικά πράγματα στα όσα ακούσαμε από του προλαλήσαντε. Πρώτα-πρώτα νομίζω ότι υπάρχει προστιθέμενη αξία που μπορεί να μας την προσφέρει το σύστημα έντες. Και όπως είπαμε προηγουμένως, η θεωρία μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ίσως έτσι το κόστος των ασφαλίστρων και ανθεκτικότητα θα βελτιωθούν και θα βελτιωθεί και η ανθεκτικότητα όλου του συστήματος. Αυτό όμως είναι ένα σενάριο. Για να ισχύσει χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται. Πέντε προϋποθέσεις έχω υπόψη μου. Να σας τις πω. Πρώτα-πρώτα για να έχει νόημα το έντες είναι να υπάρξει συνένεση για τον στόχο του συστήματος έντες. Να κρυθεί δηλαδή δόκιμη προσπάθεια το έντες. Γιατί τα αγγλικά συστήματα δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν και συστημικές κρίσεις. Γι' αυτό σας λέω, το έντες δεν είναι απαραίτητο για μεμονωμένες περιπτώσεις πτώχευσης τραπεζών. Ούτε και με τις μεγάλες μονοστημικές κρίσεις έχουμε επομένω εδώ τρία εναλλακτικά μέτρα. Αυτά τα οποία ενδεχομένω μας οδηγήσουν στο να έχουμε ένα άλλο σύστημα πιο ανθεκτικό different financial targets. Θα δούμε τώρα πώς μπράχουν τα εθνικά συστήματα εγγύσεων διαφορετωμένους στόχους. Πρώτα πρώτα να υπάρχει δυνατότητα δανεισμού από το, από το ένα σύστημα στο άλλο και από την άλλη να δούμε πώς μπορεί να βοηθήσει ο μηχανισμός σταθεροποίησης σε περίπτωση μιας συστημικής μεγάλης κρίσης και συμφωνούν τους προελίσσαντες ότι να κάνει μια μελέτη επιπτώσεων οικονομισιών θα ζυγίσει τα υπέρ και τα κατά του τι μπορεί να γίνει από τη, με τη μία μέθοδο και τι με την άλλη, δηλαδή το έντις. Άλλη προϋπόθεση. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε σχέση με το ποιο είναι ο στόχο μα εν προκειμένου. Όπως προαναφέρει και θα πρέπει να βοηθήσουμε τι τράπεζε που κατέχουν κρατικά ομόλογα. Το έντις θα είναι πετυχημένη προσπάθεια και θα αυξήσει έτσι την αξιοπιστία του κόσμου. Οπότε ε, θα υπάρχει περισσότερη ρευστότητα γιατί οι καταθέσεις από εμπιστοσύνη θα πάνε τα, τα χρήματά τους στην τράπεζα. Οπότε, προφανώς με αυτή τη ρευστότητα θα γίνουν επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα. Γιατί μόνο έτσι μπορούν να στηρίξουν τις ε, επενδύσεις. Δεν έχουν δικά τους λεφτά. Όμως, αλλού το πάει η Τραπεζική Ένωση. Εμείς θέλουμε να υπάρξει άλλου είδου σχέση κρατών και τραπεζών. Άρα, είναι δύσκολο αυτό το διάβημα, αυτή η φάση. Τώρα το θέμα του τι θα γίνει τώρα σε εθνές επίπεδο, όπου έχουμε κάποιες ισχυρές χώρες, οι οποίες δεν θέλουν να προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο. Μήπως να προχωρήσει μόνη τη η Ευρωζώνη, αργά αλλά σταθερά. Είναι σημαντικό όμως να δούμε αυτό το μέτωπο που σας ανέφερα. Τρίτη προϋπόθεση, εναρμόνιση του δίκτυ, του ορίου, του κατοφλίου, της, ε, του, του, του αξιόχρα, της ε, αξιοπιστίας για την πτώχευση. Θα πρέπει να δούμε μέχρι ποιου ε, σημείου ή από ποιο σημείο και μετά πρέπει να ενεργοποιηθεί το έντις. Άρα θα πρέπει τα όρια, τα κατόφλια να εναρμονιστούν και να μην υπάρχει ε, διαφοροποίηση σε σχέση με το πότε ε, ενεργοποιείται το ίδιο. Όπως είπαμε προηγουμένως, ε, θα πρέπει να δούμε το ότι τα εθνικά DGS έχουν διαφορετική προστασία. Αν κανείς αγοράσει ένα σπίτι, έχει διαφορετική, διαφορετικές υποχρεώσεις από ότι για άλλο είδους συναλλαγή. Να μην οδηγηθούμε δηλαδή σε στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ μελών της Ευρωζώνης προστασία των πελατών των τραπεζών περισσότερο σε κάποιες χώρες από άλλες. Όλα αυτά βέβαια θα έχουν σχέση και με το πόσο εισφέρει και συμμετέχει η κάθε τράπεζα στο σύστημα ασφάλισης των καταθέσεων. Αυτό το risk contribution. Κατά πέμπτον. Κύριε Λάγκη, αναφέρθηκε σε αυτό. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι η ποιότητα τη εποπτεία των τραπεζών. Δεν θα πρέπει να διαφοροποιούμεθα από χώρα σε χώρα, γιατί θα πρέπει όλε οι τράπεζε να κρυφθούν από το έντε. Και η Κεντρική Τράπεζα έχει ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία, ούτω ώστε να προχωρήσει προ αυτή την κατεύθυνση. Γιατί έχουμε κάποιε τράπεζε που εποπτεύονται άμεσα και κάποιε που δεν εποπτεύονται. Άρα, είπαμε, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τι μικρότερε τράπεζε. Πώ μπορούν και αυτέ να ωφεληθούν από το ΕΡΙΣ. Αλλά θα συνεχιστεί οι προβλήματισμή. Θα συνεχιστεί ο προβληματισμό για το θα γίνει με τις μικρότερες. Πέραν λοιπόν αυτών των πέντε προποθέσεων, έχουμε και κάποια άλλα ζητήματα που να τα λάβουμε υπόψη. Να δούμε πώ θα ε, δώσουν μορφή στο ΕΡΙΣ. Πρώτα πρώτα τι γίνεται με την αντασφάλιση. Το έντις είναι ένα είδο ασφάλεια, αλλά πάντοτε υπάρχει αυτό που ονομάζεται ηθικός κίνδυνος είναι και βέβαια ζήτημα αποφάσεων των κυβερνήσεων που είναι οι αποφάσεις οικονομικού χαρακτήρα. Έχουμε μικρότερες χώρες που έχουν όμως τεράστιους τραπεζικούς κλάδους. Ίσως και για φορολογικούς λόγους. Και δεν λέω ότι εκεί το, το ρίσκο είναι μεγαλύτερο, αλλά ανάλογα με το μέγεθος του τραπεζικού κλάδου είναι και το μέγεθος του ρίσκου σε περίπτωση δηλαδή του τι ζημία θα προκύψει αν πραγματοποιηθεί το ασφαλιστικό γεγονό. Άρα υπάρχουν πολλά επιχειρήματα για το πώ η, η ευθύνη τη αποζημίωση των καταθετών θα γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Άρα τα εθνικά συστήματα ασφάλισης θα πρέπει να συνεχίσουν να ισχύουν με κατόφυλλο το μηδέν. Αλλά όταν επομένω εξαντληθούν τα όρια των εθνικών συστημάτων, τότε τότε καταφεύγουμε για τα υπόλοιπα στο έντις. Συμφωνώ για το μοντέλο της αντασφάλισης που είπατε ή της αυτασφάλισης και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει επάρκεια της κάλυψης του κινδύνου. Άρα είναι θέμα πολιτικής των κρατών μελών που δεν μπορεί να χαραχθεί εκ των προτέρων. Έχουμε άλλωστε και διαφορετικά είδη κάλυψη ανάλογα με το πώ θα μεταφερθεί στο ιστορικό δίκαιο το έντες, σχετική οδηγία δηλαδή. Παρακαλώ ολοκληρώστε λέει ο πρόεδρο γιατί φτάσατε στα χρονικά όρια που έχετε ο Άρα το θέμα είναι τι σενάριο θα πρετανεύσει σε περίπτωση μεγάλης θεμική κρίση. Κάτι το έντες δεν χρειάζεται για μεμονωμένε περιπτώσει πτώχευσης και για περιπτώσεις μεγάλης κρίσης. Όμως το έντις μπορεί να συγκρατήσει το ασφαλιστικό κόστος και να αυξήσει την σταθερότητα. Όμως πρέπει να πέντε προθέσεις που ανέφερα. Ο πρόεδρος λέει ορογλώστο, ορογλώστο και άρα θα πρέπει να δούμε την κατανομή της ευθύνη σε εθνικό επίπεδο. Γι' αυτό και δεν νομίζω το άρθρο 114 θα μας προστατεύσει για την στρέψη ανταγωνισμού μεταξύ των διαφορετικών κρατών μέλων. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Με μια κάπως διαφορετική άποψη, ο κύριος Χόφμαν από την Γερμανική Ένωση ε, Συνεταιριστικών Τραπεζών. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση αυτή. Πιστεύω ότι υπάρχουν και κάποια, ε, πρέπει να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ των διαδικαστικών βημάτων που πρέπει να κάνουμε και να το διαχωρίσουμε αυτό με τις ε, ουσιαστικές προϋποθέσεις. Για μένα είναι απαραίτητη μια σωστή ανάλυση αντικτύπου για το ευρωπαϊκό σύστημα αγγείας καταθέσεων. Χωρίς σωστή τέτοια ανάλυση δεν μπορούμε να καταλήξουμε ότι είναι το καλύτερο αυτό το σύστημα. Αν υπάρχουν λοιπόν μεγάλοι τοπικοί κλειδανισμοί και είναι απαραίτητο να υπάρξει μια ένεση ρευστότητος, υπάρχουν και άλλες ε, λύσεις εναλλακτικέ πέραν του ίδις. Μπορούν να υπάρχουν ε, διευκολύνσεις για δανεισμό ή μπορεί να υπάρχουν δυνατότητες ε, ε, δανεισμού με επιστροφή. Όταν μιλάω λοιπόν για μια ανάλυση αντικτύπου, η ανάλυση αυτή θα πρέπει να σκεφτεί περισσότερο και για το πώς λειτουργεί το τωρινό σύστημα εγγύησης καταθέσεων όταν όλα τα κράτη έχουν εφαρμόσει αυτά που προβλέπονται από την νομοθεσία και έχουμε κάποια εμπειρία με αυτή την εφαρμογή για κάποια χρόνια ώστε να μπορούμε να τα αναλύσουμε. Δεύτερον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γενικά βελτιωμένο πλαίσιο με την δυνατότητα του bail-in και της επίλυσης τραπεζών και την ύπαρξη του συστήματος CSM. <clears throat> Επίσης, θα πρέπει μια τέτοια ανάλυση να συγκεκριμενοποιήσει την ανάγκη για το έντις και κατά να καταδείξει ποιες θα είναι οι συνέπειες οι οποίες θα προκύψουν από αυτό το σύστημα. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη και τον ηθικό κίνδυνο και τον ανταγωνισμό μεταξύ τραπεζών μέσα και εκτός της ζώνης του ευρώ. Θα πρέπει να αναλύσουμε το κόστος και την χρηματοδότηση ενός επιμερισμένου συστήματος εγγύησης καταθέσεων και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ο, να εξετάσουμε και τον αντίκτυπο στα λεγόμενα θεσμικά συστήματα προστασίας. Για μένα μια τέτοια ανάλυση θα πρέπει να ακολουθηθεί από μια δημόσια διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους, κάτι το οποίο δεν ελέγχθη μέχρι τώρα. Έρχομαι τώρα στα πια ουσιαστικά, ουσιαστικά θέματα. Το θέμα του ειδικού κινδυνού λόγω της μεγάλης διαφοράς σε επικινδυνότητα των εθνικών συστημάτων τρα, τραπεζικού χαρακτήρα. Αυτή η διαφορά δεν μπορεί να καλυφθεί από μόνο τιμολόγηση ή από Συμβολέ που βασίζονται στον κίνδυνο. Αυτό αρέσει σε πολλού, αλλά είναι πολύ μεγάλη οι διαφορέ για να μπορέσει να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστημα. Δεν είναι μόνο θέμα μεγέθου όπω αναφέρθηκε προηγουμένω. Οι κίνδυνοι στις, ε, ε, στο ευρωπαϊκό σύστημα θα πρέπει να μειωθούν ώστε να έχουμε πραγματικό επιδε, ε, επιμερισμό. Υπάρχει η επικέντρωση στο κρατικό χρέο, υπάρχουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια πρέπει να ληφθούν υπόψη και πρέπει να υπάρξει επίση και μία επιθεώρηση μια, της ε, αξίας των στοιχείων ενεργητικού για όλες τις τράπεζες και όχι μόνο συστημικά σημαντικές τράπεζες για να μπορέσει να καταλάβει κανεί τον κίνδυνο σε τράπεζες και τα εθνικά συστήματα. Το τρίτο σημείο είναι ακριβώς αυτό που είπαμε, την αποσύνδεση των τραπεζών από το κρατικό χρέος. Εδώ θα τόνιζα ότι θα πρέπει να υπάρξει στάθμιση κινδύνου για το εθνικό χρέος και ένα όριο στην συγκέντρωσή του στα χαρτοφυλάκια. Αλλιώ τα τοπικά, τοπικοί κλειδονισμοί που γίνονται από μια ασθενική, από ασθενή ε, κρατικά ομόλογα μπορούν να διοχετευθούν στο συνολικό σύστημα. Τέταρτον, θα πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση του πτωχευτικού δικαίου και των διαδικασιών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σαφές ότι μπορούμε να έχουμε διαφορές διαδικαστικά στοιχεία στην ιεραρχία των πιστωτών στο πώς θα μπορέσει να υπάρξει αν υπάρχει μια διαφορά λοιπόν στην μεταχείριση των πιστωτών, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγάλη αβεβαιότητα γιατί θα υπάρχουν διαφορετικές επιπτώσεις χωρίς ένα κοινό σύστημα. Πέμπτο στοιχείο και είναι αυτό ουσιαστικό και πάλι, υπάρχουν δυνατότητες να υπάρχουν εναλλακτικά μέσα και συστήματα προστασίας των ε, καταθετών. Θα πρέπει να έχουν θέση σε οποιοδήποτε σύστημα, γιατί έχουν καταδείξει και την αξία τους. Η πρόταση για το ΕΝΤΙΣ είναι πάρα πολύ αρνητική και δημιουργεί προβλήματα για τα θεσμικά συστήματα προστασίας και τα αναλλακτικά συστήματα, παρά το γεγονός ότι τα συστήματα αυτά έχουν μόλις αναγνωριστεί πρόσφατα αυτά τα συστήματα. Πολλοί έχουν κάνει μία ε, σύγκριση με το αμερικάνικο σύστημα, το FDIC, Μπορώ να σας πω όμως ότι οι γερμανικές ε, συνεργατικές τράπεζες δεν έχουν πάρει ποτέ χρήματα από τους καταναλωτές γιατί τα συστήματά τους έχουν δουλέψει χωρίς κανένα πρόβλημα εδώ και 82 χρόνια. Είναι εξίσου λοιπόν καλό αυτό το σύστημα με το σύστημα FDIC και το ε, η πρόταση για το EDS έχει δημιουργήσει μεγάλη δυσπιστία και ανησυχία μεταξύ των μελών και των πελατών των συνεργατικών μας τραπεζών. Και αυτό ισχύει και για άλλες τραπεζές τέτοιου χαρακτήρα σε άλλα κράτη-μέλη. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η νομοθεσία των ε, Βρυξελών δεν πρέπει να καταστρέψει τα θεσμικά συστήματα προστασία που ήταν πάρα πολύ θετικά για να μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, την προστασία των ε, ε, καταθετών των οικονομιών μας. Και τέλος, οι Ευρωπαίοι πολίτες όλα τα κάτι μέλη θα πρέπει να καθισχαστούν ότι ένα τέτοιο σύστημα θα δώσει μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας και δεν θα οδηγήσει σε μία όχι ισοδίκαια μορφή επιμερισμού κινδύνων. Η πρόταση τώρα όπως έχει δεν πρόκειται να κερδίσει τις καρδιές πολλών Ευρωπαίων πολιτών θα ήταν επικίνδυνο να προχωρήσει κανείς με ένα τέτοιο σύστημα και να παραγνωρίσει τις πραγματικές ανησυχίες που νιώθουν οι πολίτες και οι ψηφοφόροι σε πολλά κράτη-μέλη. Γι' αυτό χρειάζεται μια πολιτική, μια διαδικασία διαφάνειας και να εξετάσουμε και όλες τις εναλλακτικές δυνατότητες επίσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία... Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, εμείς στηρίζουμε πλήρως την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συμφωνούμε με την πρόταση για ένα τελείως αμοιβαιοποιημένο σύστημα μέχρι το 2024. Νομίζω όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αν είναι να έχουμε μια τραπεζική ένωση γιατί έτσι θα υπάρχει λιγότερη σταθερότητα, θα βελτιωθούν οι μηχανισμοί μετάδοσης νομισματικής πολιτικής και θα αποφευθεί ο κατακαιρματισμός της αγοράς. Για να υπάρχει μια πραγματική τραπεζική ένωση πάντα μιλάμε για τρεις πυλώνες. Αυτός είναι ο τρίτος πυλώνας. Έχουμε δηλαδή ένα κοινό υποπτικό πλαίσιο ήδη το οποίο θα μειώσει τις πιθανότητες χρεοκοπίας τραπεζών. Έχουμε ένα κοινό πλαίσιο ε, που θα ελαχιστοποιήσει το κόστος ε, και αυτό το οποίο χρειάζεται ακόμα άρα είναι ένα μέσο για να μοιραζόμαστε τον κίνδυνο. Έχουμε δύο ε, που μειώνουν τον κίνδυνο και υπάρχει, χρειαζόμαστε αυτό το οποίο θα μας κάνει να μοιραστούμε τον κίνδυνο. Δεν είναι αφηρημένη η συζήτηση. Νομίζω πως σε μια νομισματική ένωση είναι απολύτως λογικό να υπάρχει ένα αμοιβαιοποιημένο σύστημα εγγύησης ε, καταθέσεων. Το θέμα είναι λοιπόν πώς θα προλάβουμε αυτά τα οποία αναφέραμε περίεργα κίνητρα, ηθικός κίνδυνος ή έλλειψη χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Νομίζω πως ε, κατά την απόψή μας η σταδιακή προσέγγιση της Κομισιόν είναι οπωσδήποτε σωστή. Είναι λογικό να προχωρήσουμε βήμα-βήμα και να ξεκινήσουμε με τις φάσεις ε, ασφάλισης ε, και συνασφάλισης. Αν λοιπόν υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία ε, είναι εξίσου σημαντικά δεν πρέπει να καθυστερήσουν. Δεν πρέπει δηλαδή να καθυστερήσει ο τρίτος πυλώνας όπως δεν καθυστέρησαν και οι δύο πρώτοι. Έχουμε λοιπόν μια τραπεζική ένωση χωρίς πολλά από τα πράγματα τα οποία λέγαμε. Έχουμε τους δύο πρώτους πυλώνες χωρίς ε, ενιαίους ε, χωρίς ενιαίο πτωχευτικό δίκαιο. Στις ΙΠΑ επίσης υπάρχει τραπεζική ένωση χωρίς ε, ενιαίο πτωχευτικό δίκαιο. Υπάρχει λοιπόν κάποιο προηγούμενο τώρα. Τι θεωρούμε ότι είναι, ποια βήματα είναι αναγκαία. Τρία θεωρώ. Πρώτον, για να προωθηθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα χρειάζεται τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν την οδηγία για την εγγύηση των καταθέσεων. Έτσι θα έχουμε ε, ίσους όρους ανταγωνισμού αλλά οπωσδήποτε δεν θα πρέπει να αποτελέσει τροχοπέδι για να προχωρήσει το σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Πρέπει να είναι σαφές πως η απλή εναρμόνιση των εθνικών συστημάτων δεν επαρκεί για να έχουμε μια ενιαία τραπεζική αγορά. Όσο η αποτελεσματική προστασία των καταθέσεων συνδέεται με την φερεγγιότητα ενός κράτους οι καταθέτες δεν θα εξετάζουν καθόλου τον ισολογισμό της τράπεζας αλλά την έδρα της μόνο. Δεύτερον, για το θέμα του ηθικού κινδύνου θεωρούμε πως οπωσδήποτε χρειάζονται κάποιες εισφορές ε, που θα βασίζονται στον κίνδυνο για να ε, χρηματοδοτηθεί σωστά το σύστημα εγγύης καταθέσεων. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια ευρωπαϊκή μεθολογία που θα την διαχειριζόμαστε κεντρικά. Θα πρέπει λοιπόν οι εισφορές της κάθε τράπεζας να σχετίζονται με τον κίνδυνο της σε σχέση με τις άλλες. Και βεβαίως έτσι θα αποφευχθεί ο ηθικός κίνδυνος. Τρίτον, για να μην υπάρχει κατακρεματισμός αγοράς θα πρέπει να υπάρχει ένα δημοσιονομικό ένας ε, δημοσιονομικός, ε, ένα δημοσιονομικό αποθεματικό. Υπάρχουν λοιπόν σχετικές ε, πρωτοβουλίες και βεβαίως για μια τράπεζα όπως εμείς πιθανώς να είναι προτιμητέο το bail από μια διάσωση. Βεβαίως απουσία όπως είπαμε ενός τέτοιου αποθεματικού υπάρχει ο κίνδυνος οι εθνικές αρχές να, να χρειαστεί να στηρίξουν τις ε, τράπεζες ε, οι οποίες βρίσκονται στην επικράτειά τους. Και βεβαίως θα υπάρχει και πρόβλημα με την ρευστότητα όπως είδαμε στο παρελθόν. Και βεβαίως υπάρχουν και άλλα βήματα τα οποία θα μπορούσαν να είναι θετικά και τα ανέφεραν συνάδελφοι όπως η εναρμόνιση του πτωχευτικού δικαίου ή τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αυτά θα μπορούσαν να είναι θετικά, αλλά δεν θεωρούμε πως θα πρέπει να είναι δικαιολογία για να καθαιρεί ο τρίτος πυλώνας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο πρόεδρος. Ο κύριος Ερίκος Μίλσεν από την Unicredit. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε. Θα ήθελα να σας τονίσω ότι είμαι ερευνητής από την Unicredit. Μιλώ ως Ευρωπαίος οικονομολόγος και όχι ως ε, εκπρόσωπος μιας τράπεζας. Ελπίζω ότι θα μπορέσετε να το αναγνωρίσετε αυτό. Εγώ υποστηρίζω το Ίντις ως τον ελίποντα κρίκο ή τον τελευταίο κρίκο στην Τραπεζική Ένωση και αυτό είναι πολύ σημαντικό για πολλούς ε, λόγους. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολλά τεχνικά ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί και φυσικά θα πρέπει να τα λάβει κανείς όλα αυτά τα θέματα. Εδώ το θέμα όμως δεν είναι να δημιουργήσουμε την τελεότητα, αλλά να φτιάξουμε κάτι καλύτερο από το σύστημα που έχουμε τώρα. Λοιπόν, θα ήθελα επομένω να υπογραμμίσω μερικά θεμελιώδη θέματα που καταδεικνύουν πού βρισκόμαστε. Πρώτα απ' όλα υπάρχει η ανισομέρεια μεταξύ μιας κοινή προσέγγισης όπως λέγανε οι Αμερικανοί δεν μπορείτε να έχετε φορολογία χωρίς εκπροσώψη στην Ευρώπη δεν μπορεί να έχετε επιμερισμό κινδύνου χωρίς πολιτική ένωση. Ούτε όμως και το τούμπαλι δεν μπορείτε να έχετε. Να έχετε μια κεντρική αρχή και εθνική ε, ανάληψη κινδύνου. Αυτό έχουμε αυτή τη στιγμή. Αν πάρουμε μια χώρα όπως η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία, όπου υπάρχει υποπτία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και κάτι πάει στραβά. Και πρέπει να γίνει bailout από τους καταθέτες και τελικά έρχεται η... το Μπουγιουρντή από την Φραγκφούρτη που λέει τα κάναμε θάλασσα και εσείς τώρα πρέπει να πληρώσετε. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Πρέπει να υπάρχει πραγματική εκπροσώπηση όλων στην περίπτωση που θα υπάρχει επιμερισμός κινδύνων. Επομένως, η κίνηση προς μια πιο σκοντινή, πιο μια στενή ε, ένωση θα πρέπει να συμβαδίσει με την κοινή ανάληψη κίνδυνου. Το δεύτερο στοιχείο είναι σε μια τέτοια κατάσταση όταν τα στοιχεία των ε, τραπεζών, τα στοιχεία του Μάλλον τα αξιόγραφα των τραπεζών δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο γιατί υπάρχουν διαφορετικά συστήματα εγγύηση καταθέσεων. Και δεν υπάρχει επομένω μια ενιαία αγορά σε όλα αυτά τα θέματα. Κάποιοι θεωρούν, κάποιε τράπεζε θεωρούνται πιο ασφαλεί για να καταθέτει κανεί τα χρήματα ή όχι. Είναι πολλά πράγματα που μπορεί να πει κανεί, αλλά θέλω να επανέλθω σε κάτι το οποίο αναφέρθηκε το μεγάλο θέμα του επιμερισμού κινδύνου και τη μείωση του κινδύνου που υποτίθεται ότι πρέπει προηγουμένω να επιτευχθεί. Να σα πω ότι σύμφωνα απόλυτα ότι πρέπει να πάμε προς μια κατεύθυνση που θα μειωθεί ή θα καταργηθεί τελείως η σύνδεση μεταξύ τραπεζών και κρατικού χρέους. Αυτό πρέπει να γίνει όμως μέσω της Τραπεζικής Ένωσης, να υπάρχει μια κοινή αγορά για όλες τις τράπεζες η οποία θα οδηγήσει σε μια κοινή τους αντιμετώπιση, όχι με το να δημιουργήσουμε εθνικές προστασίες για τις καταθέσεις, παραδείγματος χάρη. Αυτό που εγώ βρίσκω επικίνδυνο είναι αυτό το οποίο ελέγχθη εδώ και από το προηγούμενο πάνελ την θεσμοποίηση των κινδύνων που προέρχονται από τα κρατικά ομόλογα. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα. Και έχω εργαστεί στο Διεθνές Ομοσυμματικό Ταμείο και στην Παγκόσμια Τράπεζα με πρωτού έρθω εδώ στην Ευρώπη. Μερικά παραδείγματα. Δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ του κινδύνου του κρατικού χρέους και των άλλων υποχρεώσεων μιας κυβέρνησης. Δεν μπορεί ποτέ ένα κράτος να διαρθώσει το χρέος του χωρίς να υπάρχουν επιπτώσεις για τις άλλες υποχρεώσεις του, παραδείγματος χάρη, τις συντάξεις ε, ή την υγειονομική περιθέρωση κτλ. Δεν μπορεί λοιπόν να διαχωρίσει κανείς αυτά τα πράγματα και ιστορικά δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Δεύτερον, δεν μπορείτε να φανταστείτε ότι μπορεί να διαχωριστεί το κρατικό χρέος από τον ιδιωτικό τομέα. Πάρτε την Ιταλία που έχει το δημόσιο χρέος της που προέρχεται από διάφορους τομείς ε, της κυβέρνησης. Αλλά τα νοικοκυριά που έχουν το 60% αυτού του χρέους και, αυτέ, και αυτά εμπλέκονται σε αυτήν την περίπτωση. Δεν μπορεί κανείς να αποσυνδέσει λοιπόν το ιδιωτικό χρέος από το δημόσιο χρέος. Δεν μπορεί κανείς να θεωρεί ότι το κρατικό χρέος είναι κάτι το οποίο είναι διαφορετικό, ένα διαφορετικό σύστημα, ένα διαφορετικό χρέος. Και επίσης σκεφτείτε τα τελευταία χρόνια τι έχει γίνει με την εξαίρεση Ελλάδος που ήταν μια εξαιρετική περίπτωση. Δεν είναι το κρατικό χρέος που δημιούργησε προβλήματα για τις τράπεζες. Στην κρίση του 2008-2014 τα στοιχεία του Δούνου του λένε ότι χρειάστηκαν τα 12% του ΑΕΠ στη Γερμανία για τη διάσωση των τραπεζών. και ήταν πολύ μικρότερο το ποσοστό σε χώρες με μεγάλο χρέος όπως η Γερμανία και η Ιταλία παρόλα αυτά. Δεν υπάρχει λοιπόν σύνδεση. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, ενέκρινε ε, μια μεγάλη χρηματοδότηση για μια τράπεζα, μια τράπεζα που έχει σαν βασικούς μετόχους το κράτος του Σλέσφικ Χολστάν και του Αμβούργου τα κρατήρια αυτά στη Γερμανία. πρέπει να διαχωρίσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει μόνο ο κίνδυνος από το κρατικό α, χρέος. Αν λοιπόν τα αποσυνδέσετε τα πράγματα θα δημιουργήσετε ένα υπερκυκλικό σύστημα το οποίο δημιουργεί μεγαλύτερους κινδύνους. Με τον τρόπο αυτό εσείς κινδυνεύετε να αυξήσετε τον κίνδυνο για μια κρίση. Στι κρίσει δεν ήταν εθνικέ τράπεζε στην Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία που δημιούργησαν το πρόβλημα με την πώληση του χρέου. Ήταν οι μεγάλε ευρωπαϊκέ τράπεζε οι οποίε είχαν τρισεκατομμύρια καταθέσεων ή στοιχείων ενεργητικού στις περιφερειακές χώρες όπου υπήρξαν σημαντικέ αποσύρσεις και αυτό οδήγησε σε όξυνση της κρίσης. Θα ήθελα να σταματήσω εδώ να πω ότι είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος ε, σύνδεσης μεταξύ κρατικού χρέους και τραπεζών. Πρέπει να γίνει ε, διαχωρισμός, αλλά με διαφορετικό τρόπο και χρειάζεται το κοινό σύστημα εγγύησεων. Συμφωνώ, συμφωνώ προσωπικά. Ακριβώς αυτά τα μέτρα αναγγελίας κινδύνου. Έτσι, αυτό μου αρέσουν. Αυτά, αυτά. Τώρα ο κύριος Λούκε ζητεί τον ε, λόγο. Α, συγγνώμη. Συγγνώμη, συγγνώμη, τα μπέρδεψα. Γιατί πρώτα-πρώτα θα πρέπει να λάβουν το λόγο ε, οι, οι με το ΚΑΤΣΔΙ. Θα φύγουν οι διερμηνές και θα τα πούμε μετά στα αγγλικά, αλλά τέλος πάντων, γρήγορα, γρήγορα. Κύριε Λάγκεν, ναι, ναι, όσον αφορά ε, αυτά τα συστήματα προστασίας. Άκουσα τι είπατε. Πώς έχουν λειτουργήσει αυτά τα συστήματα σε κάποια πρώιμη φάση. Και ρωτώ, βέβαια, εσείς μας τα είπατε με πολλά ερωτηματικά σε σχέση με το κατά πόσον χρειάζεται το έντις. Αλλά αντιστρέφω το ερώτημα, στα πλαίσια του έντις Πώς θα εξασφαλίσουμε το σύστημα να λειτουργεί εύρυθμα όπως και στην αρχή, όπως γινόταν δηλαδή στην πρώιμη εκείνη φάση, αντιστρέφω το ερώτημά Τώρα, όσον αφορά τον κύριο, ε, την κυρία από την Τράπεζα Σανταντέρ, είπατε ότι η μείωση του ρίσκου δεν θα πρέπει να είναι μια πρόφαση να μην ξεκινήσουμε το έντις Οπότε, εάν ε, συνοψίσουμε αυτά που ακούσαμε σήμερα, είπαμε ότι ο καθένα εξετάζει άλλη φάση του έντε και μας λέει ότι άλλα χρειάζονται σε κάθε φάση για το σύστημα. Άρα, επενδύσω ότι χέρι-χέρι πρέπει να πάει η μείωση του κινδύνου με την κατανομή του κινδύνου. Συμφωνείτε ή όχι ότι για κάθε φάση ε, αντασφάλιση, αυτασφάλιση, συνασφάλιση θα έχουμε διαφορετικό επίπεδο μείωσης του κινδύνου. Και τι θα πρέπει να γίνει. Και τελευταίο, αλλά σημαντικό τώρα. Ο κ. Νίλσεν μας τα είπε έξω από τα δόντια για το κίνδυνο του κρατικού χρέους. Και εδώ και το ζουμί τη σημερινής συζήτησης. Μετά όλα όσα είπατε και που έχω σημειώσει εδώ, θα συμφωνούσατε με αυτά που ακούσαμε προηγουμένω για την έκθεση των τραπεζών μας στον κίνδυνο του κρατικού χρέους και άρα θα πρέπει να υπάρξει ένα όριο στο πόσο μια τράπεζα θα πρέπει να είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο κρατικής πια κρίση. Η κυρία Φερέιρα θα σας το πω πολύ σύντομα για τους δύο πρώτους. Έχω μια ακούσει τα επιχειρήματα που υπάρχουν και αυτά που μας είπατε. Και εσείς τι λέτε, αυτά τα θέματα ισχύουν, όλα αυτά που μας είπατε, τα επιχειρήματά σας ισχύουν, μια που έχουμε ήδη τους πρώτους δύο πυλώνες της ε- Τραπεζικής Ένωσης και άρα ε, θα πρέπει να αφιερωθούμε ότι όλα αυτά είναι προϋποθέσεις πριν αρχίσει ο τρίτος πυλώνας της Τραπεζικής Ένωσης γιατί θα πρέπει να υπάρξει η αυτοπεποίθηση του ΖΙΠΗΝ να προχωρήσουμε στην ευρωπαϊκή εποπτεία μια που θεωρούσαμε ότι υπάρχουν οι κοινοί κανόνες, τα μέτρα μείωσης του κινδύνου και είπαμε να έχουμε αυτόν τον ενιαίο μηχανισμό εξυγκίασης. Αλλά μετά πάει η κοινή ε, εγγύηση των καταθέσεων. Thank you. Σας ευχαριστούμε εμείς. Αυτό εμένα με κάλυψε ο οπότε δεν θα μιλήσω. Να πω πως εκτιμώ αυτό το οποίο ζήτησε ο κύριος Χόφμαν, ε, δηλαδή μια αξιολόγηση αντικτύπου και το ότι ζητήσατε και μια δημοσία διαβουλευσία. Ευχαριστώ. Σιλβί Γκουλάρ. Με συγχωρείτε που έλειπα. Σύντομα, τι άποψη έχετε για την άποψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και το ότι βεβαίω ζητάει κάποιο αποθεματικό για το ένδυση. Ο κύριος Παπαδημούλης. Ευχαριστώ. Ποια είναι η προσέγγιση σας για την διαδικασία των τριών πυλών. Όλα τα προαπαιτούμενα τα οποία έχετε θέσει για τη δημιουργία του τρίτου πυλώνα αφορούν μόνο αυτό. Είχατε και ανάλογες ε, διαφωνίες για τα προηγούμενα βήματα της διαδικασίας. Σας ευχαριστώ κύριε Λάμπερτ. Έφυγε. Κύριε Τσάνη δεν είναι εδώ. Κύριε Σάνεμανς, ναι, κύριε Πρόεδρε, έχω ένα ερώτημα. Να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές ε, και τον πρόεδρο της Επιτροπής. Ε, χαρακτηριστικό είναι βεβαίως στο τέλος να έχουμε ε, μια ακρόαση για την τελευταία φάση της διαδικασίας αυτής και δεν ξέρουμε ακόμα για το εάν ε, θα υπάρξει αυτή η διαδικασία. Οι Έλληνες φίλοι μας βεβαίως χαίρονται ιδιαίτερα, δεν βλέπουν την ώρα, η Σανταντέρ το ίδιο. Χρειάζεται λοιπόν αλληλεγγύη για αυτό το θέμα. Η αλληλεγγύη βεβαίως ε, θα πρέπει να έρχεται από τις εθνικές ε, ταυτότητες. Δεν είναι ντροπή. Οι πολιτισμικές διαφορές επίσης δεν είναι ντροπή. Μόνο έτσι, αν τα διατηρήσουμε αυτά, θα υπάρξει αλληλεγγύη. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Λούκε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι περίεργο το ότι οι δύο πρώτοι ομιλητές <coughs> ζήτησαν και διαβούλευση και μια μελέτη που ενώ η επόμενη που είναι υπέρ του Ευρωπαϊκού Συστήματος όχι. Αυτά λοιπόν τα οποία είδαμε αφορούν και πάντα μας λένε για μια για ένα θετικό αποτέλεσμα το ότι θα μοιραζόμαστε τον κίνδυνο και υπάρχει ο νόμος των μεγάλων αριθμών και βεβαίω υπάρχει και το αρνητικό ο κίνδυνος ο ηθικός, ο οποίος νομίζω είναι γεννή σε ένα σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Αν δούμε αυτό το οποίο μας λέτε για θετικό το νόμο των μεγάλων αριθμών, Πραγματι αυτό ισχύει εάν δεν υπάρχει συσχετισμός μεταξύ των ε, κινδύνων. Αλλιώς βεβαίως ο νόμος των μεγάλων αριθμών ε, δεν ισχύει τόσο πολύ. Οπότε αυτό το οποίο μας παρουσιάζεται ως θετικό ίσως να μην ισχύει τόσο. Ενώ ο ηθικός κίνδυνος είναι ισχυρότερος από ό,τι μας λέτε. Γιατί το επιχείρημα βεβαίως είναι πως θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποιο, κάποιες εισφορές με βάση τον ε, κίνδυνο. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν ακριβώς υπησέρχεται ο ηθικός ε, κίνδυνος. Στην περίπτωση των ασφαλίστρων. Έχουμε λοιπόν θετικά και αρνητικά σύμφωνα με τα όσα μας είπαν οι ομιλητές και το ερώτημά μου είναι το εξής. Δεν υπονομεί αυτό ότι θα πρέπει πρώτα να γίνει μια αξιολόγηση αντικτύπου για το ποια από αυτά τα αποτελέσματα είναι πιθανότερα. Θα είχατε δηλαδή το ίδιο συμπέρασμα με τους πρώτους ομιλητές, ότι θα πρέπει να γίνει πρώτα μια δημόσια διαβούλευση πριν λάβουμε απόφαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Παύλο Τόλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και, τους, και τα τέσσερα μέλη του πάνελ. Θέλω να πάρω την οπτική γωνία του απλού πολίτη. Μιλάμε πολλές φορές με την οπτική των χρηματοπιστωτικών ε, φορέων, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε ότι ο στόχος μας είναι να έχουμε μια τραπεζική ένωση. Ένας πολίτης όμως στην Ιταλία, στην ε, Ισπανία, δεν ενδιαφέρεται πού βρίσκεται η τράπεζα σε ποια περιοχή της Ισπανίας ή της Ιταλίας. Θα ήθελα λοιπόν ο Ευρωπαίος πολίτης να έχει την ε, ίδια ε, ασφάλεια ανεξάρτητα από το αν είναι καταθέτει σε μια γερμανική, ισπανική ή ιταλική τράπεζα. Πώς λοιπόν θα το επιτύχουμε αυτό με την ε, πρόταση του Ίντις, αυτό είναι το ερώτημά μου. Υπερβάν Σουπερές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για όλες αυτές τις παρεμβάσεις που πολλές φορές συμφωνούν, αλλού διαφέρουν. Ίσως θα έπρεπε να διοργανώσουμε και μια δεύτερη ακρόαση που να εκφραστούν και άλλες απόψεις, οι οποίες δεν μπόρεσαν να εκφραστούν σήμερα. Αλλά θα ήθελα να ζητήσω από το πάνελ να επανέλθει σε κάτι που μας είπε στο πρώτο πάνελ ο Γκούτραν Βόλφ για τους κινδύνους στρέβλωσης μεταξύ ενός συστήματος το οποίο είναι ολοκληρωμένο ως προς την εποπτεία αλλά ενός συστήματος εγγύησης καταθέσεων το οποίο παραμένει στα χέρια των κρατών μελών. Υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνος να εκτεθούν οι καταθέτες σε αποφάσεις που έχουν περάσει σε ένα πιο ψηλό ομοσπονδιακό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά και μία μεταφορά κυριαρχίας. Και δεν ξέρω αν έχουμε μετρήσει όλα τα, όλο τον αντίκτυπο που μπορεί να προέλθει. Επίσης, πριν δημιουργήσουμε το Ταμείο Εγγυήσεων, χρειάζεται μία μελέτη αντικτύπου. Μήπως λοιπόν θεωρείτε ότι θα πρέπει η διαδικασία αυτή του ελέγχου αντικτύπου και να καθυστερήσει το σύστημα ευρωπαϊκών εγγύησεων δεν θα μας εκθέσει σε περαιτέρω κινδύνους. Και τέλος να ρωτήσω τους πανελιστές, τα μέλη του πάνελ, αν θεωρούν ότι οι διατάξεις της Τραπεζικής Ένωσης όσοι έχουν σήμερα μπορούν να λειτουργήσουν. Γιατί αν πάρουμε μια κάποια απόσταση από τα πράγματα, εδώ έχουμε ένα ευρωπαϊκό θέμα. Έχουμε προχωρήσει δύο βήματα και έχουμε υπαναχωρήσει για το τρίτο βήμα. Και η ιστορία μας διδάσκει ότι κάθε φορά που το κάνουμε αυτό, κάνουμε πιο εύθραυστα τα δύο προηγούμενα βήματα που έχουμε κάνει. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από τα μέλη του πάνελ να μου πούν αν θεωρείτε ότι η πολυμερής εποπτεία είναι πρόοδος, αν θεωρείτε ότι το Ταμείο Επίλυσης είναι πρόοδος ή μήπως θεωρείτε ότι αν, ε, αν, αν θέσουμε να αφιβόλω αυτές τις δύο επιτεύξεις θα οδηγήσει και σε ένα αφόρητο κίνδυνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ βλέπω ένα μεγάλο κίνδυνο για τους δύο αυτούς πυλώνες της ε, Τραπεζικής Ένωσης αν δεν μπορέσουμε να θεσπίσουμε και το τρίτο πυλώνα πολύ σύντομα. Τελευταίος, θα είστε σύντομοι γιατί ε, τελειώνει ο χρόνος ο κύριος Χάιας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω τρία ερωτήματα. Το πρώτο είναι πολιτικό ερώτημα. Αναρωτιέμαι αν τη στιγμή που βρισκόμαστε στην κρίση το 2009 με 2011 πρότεινε κάποιος να μην έχουμε μια εγγύηση των καταθετών. Τι θα σκεφτόταν τότε, ότι δεν είναι καλή ιδέα ή ότι είναι καλή ιδέα όσο απομακρυνόμαστε από την κρίση, η ανάγκη του να έχουμε ένα τρίτο πυλώνα για την Τραπεζική Ένωση, κάτι το οποίο το δεχόμαστε όλοι, μειώνεται κάπως αυτή η επιτακτικότητα και πρέπει να θέσουμε λοιπόν αυτό το πολιτικό ερώτημα. Και το ερώτημα μου τα μέλη του πάνελ είναι το εξή. Είναι θέμα χρόνου και χρονισμού μεταξύ της ασφάλισης, της συνασφάλισης, και της πλήρους ασφάλισης. Μπορούμε να μιλήσουμε για το χρόνο με τον οποίο πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία του επιμερισμού. Είναι θέμα χρόνου όμως ή έχουν πραγματική αντίρρηση για το θέμα αυτό. Είναι πράγματι θέμα αρχών αν το δέχεστε αυτό σε βάση Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όχι. Ή τουλάχιστον ζώνης ευρώ. Και για τον κύριο Φαν Ρόσπεκ. Μιλήσατε προηγουμένως για την ποιότητα της τραπεζικής εποπτείας που είναι ο πρώτος και ο βασικός πυλώνας της ε, Τραπεζικής Ένωσης. Και επειδή κάποια τμήματα της εποπτείας θα αναφορούν τις μικρές τράπεζες, ήθελα να πει ότι αν περάσουμε σε ένα καλύτερο σύστημα, πιο πλήρες σύστημα εποπτείας των τραπεζών, όπου θα εμπλέκεται και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για όλες τις τράπεζες, αν θα συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα άλλαζε η θέση του σε σχέση με το ίδιο σε επίπεδο αρχών. Σα ευχαριστούμε εμεί κύριε ο Κύριε Φαν Ρόζιμπεκε, έχετε πρώτο το λόγο. Σα ευχαριστώ για τι ερωτήσει σα, Σας ομαδοποιήσουμε την τελευταία με την δεύτερη κυρία Σφερέρα. Όχι, δεν έχω καμία ε, κατηγορηματική αντιθέση στο Ίντις, ούτε έχω κάποιο άλλο συμφέρον να μην γίνει. Πάντω, εάν θα γίνει, θα πρέπει να γίνει 100% και να γίνει με τον ορθό τρόπο. Και τα κριτήρια τα οποία σας είπα εκτός μικροφώνου κυρία Φερέ. Um, ναι, ναι, θα σας πω, θα σας πω, λέει ο κύριος Ρόζεμπε και βεβαίω και θα λάβουμε υπόψη το δεύτερο πυλόν της Τραπεζικής Ένωσης και αυτό το έχουμε πει και ξαναπεί, επαναλαμβάνομαι ότι ξεκίνησε στραβά το πράγμα. Άρα θα πρέπει να κοιτάξουμε τι γίνεται με την Μπέι Αλίν τι γίνεται με την Μπέρντ Άρα θα πρέπει να ξαναπροβληματιστούμε. Να ε, δούμε τι έγινε το SRM. Ε, δηλαδή, το, αυτό που χρειάζεται είναι η ασφάλιση έναντι του κινδύνου. Α, επομένως, το σενάριο είναι περισσότεροι κίνδυνοι ε, και να σας πω την αλήθεια, δεν με νοιάζει αν έχουμε εθνικά συστήματα, αλλά αν έχουμε ένα ευρωπαϊκό, ένα έντις, ε, να το κάνουμε σωστά τότε. Αυτό προσπαθώ να πω. Κύριε δεν έχω κάποια κάθετη αντίθεση και δεν με νοιάζει εάν η Κεντρική Τράπεζα θα υποπτεύει τις μικρότερες. Ίσως θα ήταν καλό για το έντις, εάν ήταν δυνατόν να κοπούν αυτοί οι δεσμοί που είπαμε εθνική εποπτεία και εθνικές εποπτικές αρχές. Τώρα, άλλες ερωτήσεις δεν έπιασα το όνομά σας και από το Προεδρείο κάποιος είπε κάτι ενδιαφέρον εάν υποθέσουμε ότι αποδίδει το έντις και αναβαθμίζει την ε, εμπιστοσύνη των καταθετών σε όλη την Ευρωζώνη. Αυτό θα ήταν φανταστικό. Θα σήμαινε ότι πετύχαμε. Όμως συνεχίζει το πρόβλημα ότι έχουμε τραπέζες εκτός Ευρωζώνης που έχουν ανταγωνιστικό μειονέκτημα γιατί το σύστημα της Ευρωζώνης προσφέρει περισσότερα προστασία. Οπότε θα βρεθεί το θέμα κατά πόσο αυτέ οι άλλε τράπεζε μπορούν να μπουν στην Ευρωζώνη και να κρυφθούν από το έντις. Πολύ σημαντικά αυτά. Έχουμε και το άρθρο 1.1.4. Έτσι είπαν οι, οι νομικοί μα ότι θέλουν το 352 και όχι το 114. Να συνεχίσει αυτό να ισχύει. Όχι, να μην πάμε δηλαδή σε δια, διακυβερνητική συμφωνία. Τώρα για το θέμα του backstop και την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Τράπεζα. Τώρα δεν ισχύει το backstop για το DGS. όχι για την οδηγία αυτή του συστήματος εγγύηση καταθέσεων και είπαμε ότι δεν υπάρχει εκεί πέρα ευθύνη προς το παρόν. Και άρα δεν ξέρουμε όμως πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε σχέση με το τι θα ισχύσει στην πραγματικότητα. Άρα τα πράγματα είναι κάπως τριμωγμένα. Και τώρα ξαναγυρίζουμε στο πρώτο θέμα που σας είπα, ότι η οδηγία για το για την εγγύηση ε, δεν μας καλύπτει και ξαναγυρίζουμε στο θέμα του backstop. Άρα ό,τι σύστημα για να υπάρχει θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να καλυφθεί η ζημιά όποτε πραγματοποιηθεί το σενάριο κάποιας κρίσης που σοβεί τοπικά. Κυρία Φεραίρα